Okay. Καλώς ήρθατε όλοι. Θα συνεχίσω στα Ιταλικά τιμώντας την πολυγλωσία. Πρέπει να φορέσετε όλοι τα ακουστικά σας προς τιμήν της πολυγλωσσίας. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω όλους. Να καλωσορίσω επίσης και τους εμπειρογνώμονες και προσκεκλημένους, τους οποίους έχουμε ανάμεσά μας σήμερα. Παρακαλώ λίγη ησυχία, ξαναλέει η Πρόεδρος. Έχουμε τον καθηγητή Νίκ Σάβελ. Πολιτικές ακολουθητές και εφαρμογή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε επίσης τον κύριο Μαρτίνιουκ, διδασκαλία ξένων γλωσσών. Και ο Μικέλε Γκατζόλα, ωφέλη και στρατηγική της πολυγλωσσίας. Αυτά είναι τα τρία θέματα. Ευχαριστώ επίσης και ε, τις υπηρεσίες της επιμελητιακές της Επιτροπής μας Ζούμε μια δύσκολη στιγμή στην Ευρώπη και όχι μόνο και γύρω από το θέμα της πολυγλωσσίας. Υπάρχουν ε, γύρω από το θέμα της πολυγλωσσίας επιμέρους θέματα όπως ε, η δραστήρια προστασία της ποικιλότητα ε, της πολυγλωσσίας πρέπει να είναι χαρακτηριστικό τμήμα των πολιτικών που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον πολιτισμό. Ενθυμίστε την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής, εννοώ του 2010. Ο άλλος πυλώνας είναι η προώθηση της εκμάθησης των ξένων γλωσσών, όχι μόνο από τους νέους, αλλά κατά τη διάρκεια της ζωής τους από όλους τους πολίτες. είναι ένα δικαίωμα η εκμάθηση γλωσσών, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για αυτούς οι οποίοι φιλοξενούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές γλώσσες στην Ευρώπη ε, που θεωρούνται επίσημες ότι είναι αναγνωρισμένες γλώσσες, εθνικές γλώσσες, περιφερειακές γλώσσες, τα, η γλώσσα της Ουαλίας, τη γλώσσα της Φριζίας, το Γίντις και σε πολλές από αυτές τις γλώσσες ε, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες ε, και σε σχολικές δομές. Και γι' αυτό ακριβώς γίνονται προτάσεις ε, για την σωστή εκμάθηση όλων αυτών των γλωσσών. Ο στόχος είναι κάθε Ευρωπαίος, κάθε παιδί στην Ευρώπη μέσα από τη σχολική διαδικασία να φεύγει γνωρίζοντας φυσικά τη μητρική του γλώσσα συν δύο. Αυτή είναι η λογική. Έχετε λάβει αρκετά θα έλεγα στοιχεία ε, και τεκμηρίωση για την τεράστια δουλειά που έχουν κάνει πολλά Ινστιτούτα στην Ευρώπη σχετικά με τις προκλήσεις της πολυγλωσσίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε και σε ποιους τομείς εμείς σαν Επιτροπή Πολιτισμού μπορούμε να λειτουργήσουμε κατά κάποιο τρόπο ε, με πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδιαίτερα μετά και από τις προκλήσεις που δημιουργούνται από τη μετανάστευση. Υπάρχουν πανεπιστήμια επίσης τα οποία υποδέχονται πολλούς ξένους φοιτητές και έτσι έχουν αναπτυχθεί νέες διδακτικές μεθοδολογίες, νέες παιδαγωγικές μέθοδοι και γι' αυτό θα δώσω τον λόγο μέχρι 10 λεπτά σε κάθε ένα από τους τρεις εμπειρογνώμονες και στο τέλος μπορείτε να καταθέσετε τις ερωτήσεις σας και να καταλήξουμε σε ένα συνολικό σε μια συνολική εικόνα. Θα ξεκινήσω με τον Νίκ Σάβιλ για τις πολιτικές και την εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας παρακαλώ να κάνετε λίγη ησυχία, λέει η Πρόεδρος για τρίτη φορά. Σας καλωσορίζω. Ελπίζω να έχετε την έκθεση στην οποία αναφέρομαι. Ε, αυτά είναι τα έξι σημεία στα οποία θα σταθώ. Θα προχωρήσω αρκετά γρήγορα γιατί έχω μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μου. Ο στόχος τον οποίο είχαμε, αυτό που μας ζητήθηκε, είναι να δούμε ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική ε, τα τελευταία πέντε χρόνια, από το 2011 και μετά τμήμα του στόχου ε, είναι ε, η εξής επιμέρους, αν θέλετε, τα εξής επιμέρους πεδία, τα οποία θα σας τα παρουσιάσω πολύ ε, συνοπτικά. Η στρατηγική για την πολυγλωσία υιοθετήθηκε καταρχάς από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έτος 2008 οι στόχοι τους οποίους έθεσε στην απόφασή του το Συμβούλιο είναι αυτοί που βλέπετε αλλά τους γνωρίζετε δεν θα σας κουράσω. Στο πλαίσιο των στόχων αυτών μας ζητήθηκε να δώσουμε πέντε απαντήσεις τις οποίες ερωτήσεις τους θα σας δείξω στην τρίτη διαφάνεια θα δώσω τις απαντήσεις αυτές από πλευράς μου τουλάχιστον στο τέλος της παρουσίασής μου ε, υπό μορφή συμπερασμάτων. Οι πρόσφατες εξελίξεις από το 2011 δημιουργούν μια εικόνα όχι μόνο για το τι συμβαίνει με την πολυγλωσία στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν ε, πλαίσια τα οποία διαρκούν για πάνω από 25 χρόνια και μπορούμε να δούμε τι στόχους είχαμε θέσει και τι στόχους πετύχαμε. Έγιναν έρευνες ε, σχετικά με τα προγράμματα, αλλά ε, βασίζονται τα συμπεράσματα και στην προσωπική μου εμπλοκή, στην επαγγελματική εμπλοκή τα τελευταία χρόνια και στην Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Γλωσσικές Ικανότητες και στην συγκριτική μελέτη την οποία έκανε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία είναι πλάκιν προσωπικά. Λοιπόν, η ομιλία μου η γραπτή περιλαμβάνει από τις σελίδες 4 μέχρι 42 αναλυτικές απαντήσεις. Θα υπογραμμίσουμε όμως 8 συστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις μελλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη ερώτηση είναι ε, τα μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαμορφωθούν οι γλωσσικές πολιτικές των κρατών μελών και της ίδιας της Ένωσης. Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εκπαίδευση ε, περιορίζεται από την εφαρμογή των κανόνων της επικουρικότητας. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη με την ανοιχτή μέθοδο της συνεργασίας. Σαν αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας σήμερα υπάρχουν αρκετοί πόροι θα έλεγα, αρκετή τεκμηρίωση έτσι ώστε να επιλεγούν οι, ε, οι πιο ε, καλές πρακτικές. Βασικές συστάσεις λοιπόν τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να εκμεταλλευτούν τα μέσα τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως τα workshops που οργανώνει το ECML ή και τις διάφορες μορφές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Αυτά συνοδεύονται από λεπτομερείς ενημερώσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα ωφέλη της συγκεκριμένης ενέργειας. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνεται να κυκλοφορήσει ευρύτερα τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε πέρυσι τον μήνα Σεπτέμβριο στην Ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών στις Βρυξέλλες μετά την παρουσίαση μελετών στις οποίες πήρα μέρος και που είχαν σαν στόχο την απασχολησιμότητα των νέων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να ερευνηθούν και να εμβαθυνθούν. Είναι καθοριστικός ο χαρακτήρας τον οποίο έχουν οι γλώσσες για την ανάπτυξη τη κοινωνική. Είναι δύσκολο βέβαια να προσμετρήσει κανείς αντικειμενικά τα αποτελέσματα των πρωτοβουλειών αυτών αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των προγραμμάτων τους. Αυτό έχει σημασία θα έλεγα. Η δεύτερη ερώτηση είναι τα, μέσα τα οικονομικά. Αυτό καλύπτεται στη σελίδα 4 του εγγράφου που σας έχω μοιράσει και συμπληρώνονται στην σελίδα 5 με παραδείγματα. Είναι σαφές ότι το Erasmus Plus είναι η ναυαρχίδα των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης με ένα προϋπολογισμό 47 δις για τα 7 έτη του προγράμματος μέχρι το 2020. Πρέπει να εξυγχρονίσει το Erasmus Plus τις προσπάθειες που γίνονται στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Οι γλώσσες παίζουν λοιπόν σημαντικό ρόλο στο Erasmus Plus, διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή στα ερευνητικά αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα, λειτουργεί ε, σαν μοχλός δηλαδή. Και οι τρεις δράσεις αυτές είναι ευρύτατες, προωθούν την πολυγλωσία, την γλωσσική πολλαπλότητα και την διαβίου κατάρτιση. Και υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες, τις οποίες δεν θα αναφερθώ τώρα. Οι συστάσεις εδώ ε, που ακολουθούν είναι πρακτικού χαρακτήρα. Προώθηση λοιπόν της γλωσσικής ποικιλότητα και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ένα έγγραφο το οποίο να ε, παρουσιάζει συνοπτικά τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ε, προγραμμάτων που υπάρχουν σε λειτουργία σήμερα. Ερώτηση υπαριθμού 3. Ε, ευνοούνται οι προσπάθειες εκμάθησης των μεγάλων γλωσσών. Το θέμα είναι αν θα πρέπει να διατηρηθεί η κατεύθυνση αυτή ή να αναθεωρηθεί και προς ποια κατεύθυνση. Η ανάλυση την οποία κάνουμε εμείς δείχνει ότι δεν είναι ε, σωστή η παρατήρηση αυτή. Being recognized is one of the most valued assets of the EU τα θεσμικά όργανα προσπαθούν να στηρίξουν την διδασκαλία μιας μεγάλης ομάδας ευρωπαϊκών γλωσσών. Οι τρεις συστάσεις στην περίπτωση αυτή είναι ότι η πολλαπλότητα η γλωσσική και η πολυγλωσσία γενικότερα πρέπει να αναγνωρίσει τον ρόλο των Αγγλικών σαν λίγουα φράγκα στη διεθνή επικοινωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια σοβαρή προοπτική προς την κατεύθυνση αυτή. in Δεύτερον, υπό το φως των τελευταίων, αν θέλετε, μοντέλων μετανάστευσης κτλ θα πρέπει να διευρύνουμε το ρεπερτουάρ σε εισαγωγικά τον κατάλογο των γλωσσών στην Ευρώπη και δεν αναφέρομαι μόνο στις επίσημες γλώσσες. Ο στόχος μητρική γλώσσα συν 2 θα πρέπει να ιδωθεί εκ νέου υπό το φως των νέων γλωσσικών πραγματικοτήτων. Ερωτήσεις 4 και 5 που βλέπετε τώρα έχουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα καλύψει τις ανάγκες αυτών που τις χρησιμοποιούν, προωθώντας το περιφερειακό επίπεδο και εμπλέκοντας σχολεία, κοινότητες κτλ. Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης έχουν αναπροσδιοριστεί επί τη βάση των συμπερασμάτων από το παρελθόν και έχουν πραγματικά ενταχθεί στα πλαίσια των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Οι οδηγίες που ακολουθούν τα προγράμματα αυτά θα έλεγα είναι ιδιαίτερα αναλυτικές αναφέρονται στα έγγραφα της πολιτικής γύρω από τον τομέα αυτό και στις προσπάθειες χρηματοδότησης. Οι συστάσεις εδώ είναι απλές. Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να παρέχουν μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στις λιγότερο διαδεδομένες οργανώσεις και σχολεία που δεν καλύπτονται από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να το έχουν σαν δυνατότητα. Θα περάσω τώρα στις τελικές μου παρατηρήσεις. Συμπερασματικά, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της εκπαίδευσης είναι να διευκολύνουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Σχετικά με τις γλώσσες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο έχει πετύχει η Επιτροπή με αποτελεσματικό τρόπο συνεργαζόμενοι με τα κράτη-μέλη και παρέχοντας τις απαιτούμενες οικονομικές καλύψεις. Η εφαρμογή των γλωσσικών πολιτικών εξαρτάται φυσικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ως προς αυτό. Η στρατηγική όμως για την πολυγλωσσία ήταν χρήσιμη και είναι βασική δραστηριότητα στον τομέα της εκμάθησης γλωσσών. However, this strategy now now may need to be reviewed. Η στρατηγική αυτή πρέπει να αναθεωρηθεί μαζί με την βασική αρχή μητρική γλώσσα συν 2 να δώσουμε νέες προοπτικές σε σχέση με τις προτάσεις που ακούγονται από το 2008 και μετά, να λάβουμε επίσης το νέο πλαίσιο που δημιουργείται με τα αυξημένα μεταναστευτικά ρεύματα και τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών του 2015 που ενθαρρύνει την αναβάθμιση της γλωσσικής εκμάθησης στις σχολικές δομές. Πρέπει να καταστήσουμε λοιπόν να είναι πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες εκμάθησης γλωσσών και εκτός της τάξης. Το να μαθαίνει κανείς ξένες γλώσσες πρέπει να είναι ενσωματωμένο σε περιβάλλοντα φιλικά, δέκτικα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ου. Η αναθεώρηση των προγραμμάτων αυτών στη συνέχεια της στρατηγικής πολυγλωσσίας έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την συνέχιση και την διάδοση της προσπάθειας που έχει γίνει και πρέπει να υπάρξει περαιτέρω προσπάθεια που να λαμβάνει υπόψη τη νέα γλωσσική πραγματικότητα. Για να το πετύχουμε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τη διαδικασία και πολιτικά και οικονομικά συντονίζοντας τις δραστηριότητες των κρατών μελών σε περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο. Grazie eh, davvero, eh, grazie professor ehm, Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν ε, σας παρουσίασα καταλήλω. Είστε διευθυντή από το 2001 του ερευνητικού κέντρου στο ε, Cambridge, ε, στο κέντρο αξιολόγηση γλωσσών, που είναι το πιο διακεκριμένο σχετικό κέντρο. Ζητώ συγγνώμη που δεν σα σύστησε και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στο δεύτερο από του αμπειρογνώμονέ μα, τον Βάλτεμαρ Μαρτίνιουκ, για την ε, ε διδασκαλία της γλώσσας ε, και την εκμάθηση τη γλώσσα στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Οι στόχοι λοιπόν σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και την παρουσίαση μου αυτή είναι διτή. Η πρώτη ομάδα έχει να κάνει με μελέτες ε, περιπτώσεων για πολιτικές και πρωτοβουλίε που έχουν ληφθεί στα μεμονωμένα κράτη-μέλη για να βελτιωθούν οι ικανότητε ω προ την εκμάθηση γλωσσών, καθώ και μία αξιολόγηση των ε, επιδράσεων του των μέτρων αυτών δηλαδή και των ε, πρωτοβουλειών. Και ε, υποθέσεις και περιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ε, εκμάθηση και την δασκαλία γλωσσών. Η δεύτερη ομάδα έχει να κάνει με τη σύγκριση των καθεστώτων σύγκριση σε ό,τι αφορά την γνώσεις ε, των γλωσσών και κάποια έρευνα για την συμβατότητα. Και τέλος θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους στόχους ως προς τη στρατηγική και πώς συνδέονται με τα πορείσματα. Τα ερευνητικά ζητήματα λοιπόν τα οποία έθεσα προκειμένου να α, καταλήξω στα πορίσματά μου είναι τα εξή. Σε ό,τι αφορά πρώτο, την πρώτη ομάδα στόχων. Ετέθησε το ερώτημα κατά πόσον ε, οι μελέτες περιπτώσεων καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής. Το δεύτερο και ερώτημα, το οποίο είναι το υπαριθμό 3 στη διαφάνεια, είναι μελέτες και άλλες πηγές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγκριθούν τα συστήματα αξιολόγησης ε, γλωσσικών ικανοτήτων και πορίσματα σε σχέση με τη συγκρισιμότητα. Οι πόροι τώρα, τους οποίους μπόρεσα να εντοπίσω και εδώ θα πρέπει να διευκρινίσω ότι το να εντοπιστούν και να αναλυθούν, να αξιολογηθούν τέτοιες μελέτες περιπτώσεων και βέλτιστες πρακτικές στα κρατημέλη είναι τεράστια τεράστιο το έργο αυτό και πολύ χρονοβόρο. Θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο για να γίνει σωστή ανάλυση. Γιατί είναι τόσο μεγάλο ο αριθμό των πρωτοβουλειών που υπάρχουν. Άρα εγώ περιορίστηκα σε δύο συγκεκριμένα καθήκοντα σε ό,τι αφορά μελέτη περιπτώσεων και μελέτη πρακτικέ. Καταρχά, να εντοπίσω του πόρου με την πιο αντιπροσωπευτική συλλογή ευρωπαϊκών πολιτικών και πρωτοβουλειών σε ό,τι αφορά την εκμάθηση και τη διδασκαλία γλωσσών, ε, κατά προτίμηση εφόσον υπήρχαν σε μορφή βάσεων δεδομένων και να υπάρχει μια συνοπτική παρουσίαση. Και κατά δεύτερον, να υπάρχει μια αξιολόγηση των έργων προκειμένου να ελεγχθεί ο αντίκτυπος και η δυνατότητα μεταφοράς και υλοποίησης των πρακτικών αυτών αλλού. Και άρα κατά πόσον ε, μπορούν να αποτελούν να αποτελέσουν βέλτιστες πρακτικές. Τέσσερις βασικές λοιπόν πηγές ε, μπόρεσα να εντοπίσω, οι οποίες και πληρούν τους όρους τους οποίους σας ανέφερα. Η πρώτη ομάδα, πολύ χρήσιμη και πιο συνεκτική, αν θέλετε, για την προσωπική συλλογή τέτοιων περιπτώσεων. Περιλαμβάνεται στην ε, Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τις γλώσσες ε, για την επισήμανση γλωσσών. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μία τρίτη βάση δεδομένων επίσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, η οποία ε, δίδεται από το κέντρο Μόλαν για τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να δίνονται κίνητρα σε όσους μαθαίνουν γλώσσες. Επίσης, ε, πολύ χρήσιμο ήταν και η ε, έκθεση δραστηριοτήτων που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 σε ό,τι αφορά την ομάδα εργασία για την εκμάθηση γλωσσών. Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τις Γλώσσες αναπτύχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί μια εντυπωσιακή συλλογή 2.300 project που περιλαμβάνονται και τα οποία διατίθενται σε 24 γλώσσες, σε μία βάση δεδομένων όπου υπάρχει δυνατότητα αναζήτηση. Αυτό τι σημαίνει ότι όποιος θέλει μπορεί να κάνει αναζήτηση ανάλογα με τις προτεραιότητες του. Και θεωρώ ότι αυτό ενδεχομένως αποτελεί και την πιο πλούσια συλλογή τέτοιων δεδομένων. Κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να αποτελεί μια μόνιμη δραστηριότητα. Είναι λοιπόν η δουλειά την οποία ε, κάνει το δίκτυο NELIP, e, δίκτυο Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλειών και Project σε σχέση με τη γλώσσα. Υπάρχει λοιπόν μια βάση δεδομένων με project τέτοια, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια, τα οποία αποτελούν και πρωτοβουλίες με πολιτική σημασία στις 19 χώρες που είναι μέλη του project. Και έτσι επιλέχθησαν 227 ε, project από τις εθνικές υπηρεσίες και οι οποίες θεωρούνταν πολλά υποσχόμενες με μελέτες περιπτώσεων καθώς και 46 περιπτώσεις βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ορόσημα για την ποιότητα τη εκμάθηση γλωσσών και στις σχετικές πρωτοβουλίες. Η τρίτη βάση δεδομένων η οποία θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι αυτή την οποία παρέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει βάση του την έντρα του στο Γκράτ στην Αυστρία. Πρόκειται για μια μεγάλη βάση δεδομένων η οποία περιέχει 90 και πάνω από 90 ε, ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες για την εκμάθηση γλωσσών. Αυτό αυτή η βάση δεδομένων δίνει δυνατότητα και στα μέλη αλλά και στα μη μέλη του δικτύου να χρησιμοποιούν και να ωφεληθούν από τη βάση δεδομένων αυτών. Προκειμένου αυτά τα project να μεταφράζονται σε συγκεκριμένε υπηρεσίε. Και έτσι δεν σταματάει το project όταν ολοκληρώνεται η έρευνα. Συνεχίζει ο αντίκτυπο και παρέχει μια υπηρεσία στα κράτη-μέλη. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι κάποιες από τις ε, υπηρεσίες πλέον παρέχονται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τους άλλους στόχους τώρα, τα θέματα συγκρισιμότητα των συστημάτων αξιολόγηση. Υπάρχουν αρκετά τέτοια συστήματα τέσσερα τα οποία θα έπρεπε να τονίσουμε. Καταρχάς, η έρευνα τη εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τι γλώσσε, τι οποίε περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2013. Κατά δεύτερον, ε, η συγκριτική ανάλυση σε ό,τι αφορά τι γλώσσε στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση. Αναχώρα το 2014. Η επισκόπηση των εθνικών συστημάτων τεστ στην Ευρώπη, στις χώρες στην Ευρώπη. 2014 και 2015 και εδώ λοιπόν αποτελ... έχουμε μια άλλη σημαντική πηγή πόρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα βασικά πορίσματα, εξετάζοντας τις μέρες περιπτώσεων και τις βέλτιστες πρακτικές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σίγουρα υπάρχουν διάφορε πηγέ οι οποίε μπορούν να χρησιμοποιηθούν προ το σκοπό αυτό. Κάποιε είναι πολύ καλά οργανωμένες, με εύκολη πρόσβαση, με δυνατότητα αναζήτηση ε, και με μορφή βάσης δεδομένων. Ωστόσο, ο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν ελαμβάνεται απαραίτητα υπόψη όταν παρουσιάζεται το project στη φάση της παρουσίασης. Δηλαδή παρουσιάζουμε ένα project, αλλά δεν ε, υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για τη μακροπρόθεσμο αντικτύπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα μεταφορά των project, και αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση. Το project Nelly κατέληξε στο πόρισμα αυτό, στο συμπέρασμα αυτό, ότι το, η δυνατότητα μεταφοράς είναι μάλλον περιορισμένη. Γιατί η προσδοκία των συντονιστών πολλά προγραμμάτων για την ε, δυνατότητα διεθνικής ε, και διασυνοριακή συνεργασίας δεν ε, υλοποιήθηκε. Άρα σπάνια υπάρχει αυτό, αυτός ο παράγοντας της μεταφοράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκρισιμότητα των συστημάτων αξιολόγησης, αυτό περιλαμβάνεται και στι μελέτες που σας ανέφερα και έχουν γίνει πολλές τέτοιες μελέτες τα τελευταία χρόνια και τέτοιε έρευνες και συχνά μας δίνουν πολύ χρήσιμα στοιχεία και το βασικό πόρισμα είναι ότι η σύγκριση των εθνικών συστημάτων δεν είναι κάτι το ξεκάθαρο. Υπάρχει προφανώς μεγάλη διαφοροποίηση των συστημάτων και υπάρχει και μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά την ποιότητα των συστημάτων αυτών. Και εδώ νομίζω ότι το θέμα της ποιότητας προέχει της συγκρισιμότητας. Οι συστάσεις που θα μπορούσα να κάνω βάσει των ευρημάτων μου, των πορισμάτων μου, είναι οι εξή. Καταρχάς, να υπάρχει μεγαλύτερη χρήση των ήδη υφιστάμενων ε, στοιχείων και να υποστηριχθούν αυτά. Να εγκριθούν μέτρα για να υπάρχει συστηματική συλλογή και χρήση των στοιχείων αυτών και το δίκτυο NELIC για παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσε να αναδειχθεί σε μια μόνιμη διαδικασία, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο πλέον να γνωρίζουμε ότι πλέον περιλαμβάνει από 1600 στο παρελθόν 2400 τέτοια project. Επίσης, να ε, υπάρχει δυνατότητα μεταφορά των πιο επιτυχημένων προγραμμάτων, να δίνονται κίνητρα για μέτρα υλοποίησης ε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να αυξηθεί και η ποιότητα και να υπάρχουν σε όλες ε, τις χώρες συστήματα αρρωγής. Η σύσταση επίση την οποία θα ήθελα να κάνω σε ό,τι αφορά τη συνεργασία η οποία ξεκίνησε να αναπτύσσεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ήταν να συνεχιστεί η δραστηριότητα αυτή και να βελτιωθεί, να αναβαθμιστεί. Να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών προς τα κράτη-μέλη και βασικά την παροχή συμβουλών προκειμένου η υλοποίηση να μην παραμείνει ε, στην τύχη της, να υπάρχει ένα σύστημα για την υλοποίηση αυτή, καθώς και να υπάρχουν συστήματα και μελέτες για να αξιολογείται και να εκτιμάται ο αντίκτυπος για όλα τα προγράμματα που α, υποστηρίζονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you so much. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καθηγητά, μάθαμε ένα μάθημα ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν ε, κάνουμε αρκετά. Πρέπει να κάνουμε κάτι εν τέλει. Μπορεί να έχετε κάποια πρόταση από αυτό. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. των εργαλείων και των ερευνών που έχουμε. Και τώρα ο λόγος του Μικέλε Γκατζόλα, ο οποίος είναι υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Πολυγλωσία είναι από το τμήμα της εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου του Χάμπολτ στο Βερολίνο. Ασχολείται ιδιαίτερα με ερευνητικά προγράμματα ε, και ξέχασα να αναφέρω και ζητώ συγγνώμη ότι ο, ο κύριος Μαρτίνιουκ ήταν πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις Σύγχρονες Γλώσσες. Συγγνώμη που δεν το ανέφερα προηγουμένως, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρακαλώ, ε, καθηγητά Γκατζόλα. Καλημέρα, θα μιλήσω Ιταλικά, επομένως σας αφήνω λίγο χρόνο να φορέσετε ακουστικά αν τα χρειάζεστε. Λοιπόν, αντικείμενο αυτής της παρουσίασης ε, ήταν κάτι το αδύνατο τρόπον την ανέφικτο να αξιολογήσουμε το κόστος και το όφελος μια τόσο, ε, μιας τόσο ευρείας στρατηγικής όπως είναι η πολυγλωσία στην Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς ε, χρειάστηκε τρόπον την να κάνουμε κάποιες απλοποιήσεις ε, τις οποίες θα σας παρουσιάσω τώρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ε, ποια είναι τα τρία βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Πολυγνωσία. Πρόκειται για τρεις ε, στόχους, οι οποίοι είναι κοινωνικο-οικονομικοί. Ο πρώτος είναι να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και την ένταξη. Ο δεύτερος είναι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 λίγο πιο στην οικονομική σκοπιά, να προωθήσουμε την κινητικότητα στην ενιαία αγορά και στην ε, απασχολησιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και ο τρίτος στόχος, ο οποίος στην πραγματικότητα ε, κρύβεται στα συμπεράσματα και στα τελικές ε, συστάσεις, είναι να διαχειριστούμε με αποτελεσματικό τρόπο την πολυγλωσία στην Ευρώπη και να περιλαμβάνονται οι πάντες. Οι άλλοι στόχοι, δηλαδή η προώθηση της εκμάθησης των γλωσσών και να υποστηρίξουμε την μετάφραση και τη διερμηνία, είναι βασικοί στόχοι προκειμένου να επιτύχουμε τους πιο γενικούς στόχους της στρατηγικής. Όπως θα διαπιστώσετε πρόκειται για ένα πολύ ευρύ τομέα. Αυτό προσπαθούμε να αναλύσουμε. Επομένως είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες απλοποίησεις προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να αξιολογήσουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Πολυγλωσία. Μία προσέγγιση... Ε, είναι η εξή. Καταρχά, ε, χωρίζουμε την ε, παρουσίαση σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα εξετάζουμε κατά πόσον είναι απαραίτητη η στρατηγική για την πολυγλωσία. Βάσει των εμπειρικών στοιχείων που διαθέτουμε στην ε, ε, γλωσσική οικονομία προσπαθούμε να δούμε πώς αξιολογούνται οι ξένες γλώσσες στην αγορά εργασίας, ποια είναι η παρούσα κατάσταση των γλωσσικών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων και σε ποιο βαθμό η ευρωπαϊκή στρατηγική και η ευρωπαϊκή πολιτική των δύο ξένων γλωσσών πέραν της μητρικής προσαρμόζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Διότι αν μια πολιτική ε, για τις γλώσσες δεν είναι η κατάλληλη ε, για το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται, τότε δεν είναι και ε, η αρμόζουσα. Επομένως, στο δεύτερο τμήμα εξετάζουμε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον μέχρι του σημείου που διαθέτουμε στοιχεία, προκειμένου να εφαρμόσει αυτή την πολυγλωσία και να υλοποιήσει την πολιτική πολιτική που αποφασίστηκε από το Συμβούλιο. Ο πρώτο λοιπόν μεγάλο στόχο ε, που είναι οικονομικό για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Πολυγλωσία είναι κατ' ουσίαν να ευνοήσουμε μέσω τη εκμάθηση ξένων γλωσσών και άλλων μέσων ε, την απασχολησιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό το οποίο διαθέτουμε εμεί σήμερα δεν θα ήθελα τώρα να επισέλθω στις ε, ανιαρές λεπτομέρειες, μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε αναφορά θέλετε στην έκθεση είναι ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν λίγες εμπειρικές μελέτες για την οικονομική επιρροή των γλωσσών στην Ευρώπη και αυτές που έχουμε πολύ συχνά αφορούν χώρες που δεν είναι ευρωπαϊκές, όπως για παράδειγμα η Ελβετία και η Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αυξήσουμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό το οποίο διαθέτουμε και ε, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, γιατί συνήθως μαγειρεύουμε με ό,τι υλικά διαθέτουμε, είναι να δούμε κατά πόσον οι ξένες γλώσσε έχουν κάποια θετική επιρροή και στην εφημερία των ε, ε, ανθρώπων, δημιουργώντας μια καλύτερη θέση εργασία ε, και στα ωφέλη για την κοινωνία, αν έχουμε υψηλότερα στα απασχόληση και ούτω καθεξής και αν επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη. Αυτά όμω δεν είναι γενικά συμπεράσματα, ισχύουν για κάποιες χώρες για τις οποίες έχουν γίνει και σχετικές αναλύσεις. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι η γνώση της αγγλικής γλώσσας έχει ε, σαφή επιρροή στη χώρα που αναλύεται, αλλά όχι μόνο σε αυτή τη γλώσσα. Σε κάποια άλλα πλαίσια και η γνώση άλλων γνωσών μπορεί να έχει πολύ πιο σημαντικά ωφέλη από την γνώση της αγγλικής και μόνο. Ε, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Όσον αφορά την αποσχολητισιμότητα που πρόκειται για νεολογισμό που έχει προέρθει από τον αγγλικό όρο employability, ε, έχουμε κάποια προκαταρκτικά στοιχεία από μια έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερε ε, ενδείξει και άρα χρειαζόμαστε περισσότερε μελέτε. Θα προχωρήσω πολύ σύντομα αυτό που ε, προκύπτει από τις συστάσεις είναι το εξής, ότι ναι, έχουμε στοιχεία που μας δείχνουν ότι ξένες γλώσσες έχουν ωφέλη και για το άτομο ως οντότητα, αλλά και ε, συνολικά για την κοινωνία, αλλά χρειαζόμαστε καλύτερα στοιχεία για να τα αξιολογήσουμε αυτά και να αξιολογήσουμε πιο αναλυτικά τα οικονομικά ωφέλη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Πολυγλωσία. Δεύτερος γενικός στόχος είναι ο στόχος που αφορά την κοινωνική ένταξη, και την κοινωνική συνοχή και την αφομοίωση και των μεταναστών. Εδώ, ε, κατ' ουσίαν, στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει μία μεγάλη ένταση μεταξύ δύο μεγάλων μεταβλητών. Το ένα είναι η κινητικότητα, το γεγονός ότι οι άνθρωποι κυκλοφορούν ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη και από το άλλο είναι η ένταξη. Δηλαδή, ε, να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο κάποιος θεωρεί ότι συμμετέχει σε κάτι μεγαλύτερο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δικαίως θέλουν να αποφύγουν να ε, αναδυθούν στην Ευρώπη οι λεγόμενες παράλληλες κοινότητες, δηλαδή γκέτο και ξεχωριστές κοινωνίες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ευνοήσουμε την κινητικότητα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αν η παρούσα γλωσσική πολιτική που προωθείται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Πολυγλωσσία προωθεί ή όχι αυτόν τον στόχο. Η απάντηση είναι ότι μάλλον το κάνει μόνο εν μέρη. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε το 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2018 για το θέμα αυτό. Υπάρχουν διάφοροι ερευνητέ που μελετούν το ζήτημα ε, και να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα. Εδώ όμω θα σταθώ σε κάποια ουσιαστικά στοιχεία. Πρώτον, ούτε η ε, γλωσσική, πολιτική, μητρική γλώσσα και δύο ξένες γλώσσες, ούτε η γενικότερη στρατηγική επαρκούν ε, για να ε, μειώσουμε τις εντάσεις μεταξύ κινητικότητας και ένταξης. Πρέπει να δούμε τα απτά στοιχεία. Μόνο το 1 τέταρτο των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνει ότι γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες πέραν της μητρικής του και μάλιστα συνήθως είναι βασικές ή ε, ε, ενδιάμεσες οι γνώσεις που έχουμε. είναι ένα βασικό επίπεδο. Αυτά δεν θα αλλάξουν πολύ εύκολα γιατί οι Ευρωπαίοι είναι αποτελεσματικοί μέχρι ενό σημείου. Είναι πολύ δύσκολο να διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες σε αυξημένο επίπεδο. Όσον αφορά αφορά τη γνώση τη αγγλικής γλώσσα μόνο ένα 7% των Ευρωπαίων πολιτών ε, δηλώνει ότι γνωρίζει αγγλικά πάρα πολύ καλά. Οι περισσότεροι γνωρίζουν σε βασικό ή μέτριο επίπεδο μια γλώσσα, τη γλώσσα την αγγλική ε, προκειμένου. Όταν ε, ένα παιδί διδάσκεται ξένε γλώσσε στο σχολείο, δεν ξέρει ποιε γλώσσε θα του χρησιμεύσουν όταν θα γίνει ενήλικα και ποιε γλώσσε θα του χρειαστούν όταν θα θελήσει να μετακομίσει σε μια άλλη χώρα η γνώση της αγγλικής γλώσσας ως γλώσσα όχημα θα μπορούσε να βοηθήσει στην ένταξη σε μια ξένη κοινωνία, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να προλάβει την ανάδυση ε, παράλληλων, γνωσό, ε, παράλληλων κοινωνιών, διότι πρέπει να γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας στην οποία διαμένει κάποιος. Επομένως, ε, μπορούμε να έχουμε εκμάθηση της γλώσσας ε, αναζήτηση. Ε, όποιος αποφασίσει να μετακομίσει, όποιος αποφασίσει να ενταχθεί σε μια κοινότητα, θα πρέπει να μπορέσει να μάθει τη γλώσσα πριν μετακομίσει σε μια νέα χώρα και θα πρέπει να τη μάθει αμέσως μετά την άφηξή του. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα στοιχεία και αυτά είναι τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Εδώ υπάρχει ένα λάθος στη διαφάνεια. Το ε, μητρική γλώσσα συν δύο δεν επαρκεί, λείπει ένα νότεδο. Επίσης, χρειαζόμαστε περισσότερες ε, δημόσιες υπηρεσίες ε, πολύγλωσσες. Εδώ είναι πολύ σημαντική μετάφραση να μπορέσουν να υπάρχουν διοικητικά έγγραφα σε διάφορε γλώσσε. Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Ο τρίτο στόχο, έχω άλλε δύο διαφάνειε, θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου και να είμαι στην ώρα μου. Αυτό λοιπόν που σας έλεγα είναι ότι αυτός ο τρίτος στόχος υφέρπει. θέλουμε να έχουμε μια γλωσσική δημοκρατία, δηλαδή ε, μια επικοινωνία που να περιλαμβάνει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό ε, σε πολλά πράγματα. Ε, οι στοσελίδε μια γενική διεύθυνση ε, στι 3 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατίθενταν ε, σε μία μόνο γλώσσα το 2014. Οχτώ ήταν σε γαλλικά και γερμανικά και ελάχιστε ήταν διαθέσιμε σε όλες τις γλώσσες Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν μόνο την αγγλική ή μόνο αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά στην επικοινωνία του έξωθεν. Δεν αναφέρομαι στα επίσημα έγγραφα, αλλά περισσότερο στην επικοινωνία του μέσω διαδικτύου το 50% περίπου των πολιτών δεν μιλά αγγλικά, επομένως αποκλείεται από την επικοινωνία. Όσοι μιλούν αγγλικά σήμερα με ευχέρεια ή είναι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι πάνω από το 20%. Επομένως το 80% των πολιτών είτε δεν καταλαβαίνει το περιεχόμενο ή δυσκολεύεται να το κατανοήσει. Με τρεις γλώσσες μειώνεται το ποσοστό στο 25% και 50% αντιστοίχως. Το πιο ενδιαφέρον ίσως είναι ότι μόνον μόνο μία μειοψηφία κατανοεί, αλλά οι γλωσσικές δεξιότητες της ξένες γλώσσας συσχετίζονται στατιστικά και αυτό έχει αποδειχθεί με το κοινωνικό-οικονομικό ε, στάτους των πολιτών. Δηλαδή, αυτοί που γνωρίζουν ξένες γλώσσες είναι ε, συνήθως άτομα τα οποία είναι μορφωμένα και ε, έχουν και μια κάποια ε, οικονομική ευμάρεια. Δηλαδή, η γλώσσα ξένων γλωσσών δεν είναι μόνο κατά των πολιτών, αλλά είναι και κατά των ανθρώπων που βρίσκονται στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα επικοινωνίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά βάσει των στοιχείων που διαθέτουμε, το σενάριο μετά τον Brexit θα απαιτήσει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή προσοχή στην πολυγλωσία. Σας αφήνω να διαβάσετε και τα στοιχεία στην έκθεσή μου. Ολοκληρώνω την παρουσίαση περνώντα στο δεύτερο σκέλος που είναι μια αξιολόγηση του τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008 μέχρι το 2011 προκειμένου να εφαρμόσει τις συστάσεις του Συμβουλίου. Και εδώ ε, πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Κάποια αποτελέσματα πάρα πολύ σημαντικά ε, όντως τα είχαμε. Ξεκινάμε από τα καλά νέα, τα good news και ε, το αίτημα λοιπόν για τις γλωσσικές δεξιότητες των Ευρωπαίων, των παιδιών κυρίως, ε, ε, εκτελέστηκε, υλοποιήθηκε. Είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα λοιπόν που πρέπει να το επισημάνουμε. Πολλά πράγματα στον τομέα της μετάφρασης και της διερμηνίας υλοποιήθηκαν και μάλιστα τα εξηγήσαμε και καταλήλως. Ένα από τα προβλήματα, και εδώ με αυτό θα ολοκληρώσω, είναι ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποφάσισε να υποστηρίξει και μέσω χρηματοδότησης, μέσω του προγράμματος ε, της διαβίου μάθησης, του lifelong learning ή μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, τότε έχουμε κυρίω στοιχεία δεδομένα όσον αφορά του πόρου που επενδύθηκαν, δηλαδή για την πολιτική, αλλά δεν υπάρχουν δείκτε ω προ τα αποτελέσματα. Προκειμένου λοιπόν να μονιμοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική και να διαπιστώσουμε ότι όντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε μέσω τη άμεση συνεισφορά να υποστηρίξει την αποσχολησιμότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών, χρειαζόμαστε δεδομένα για το τελικό αποτέλεσμα αυτών των προγραμμάτων. Να δούμε αν όντω μέσω των προγραμμάτων ε, είχαμε κάποιες σημαντικές συνέπειες όσον αφορά τις ικανότητες των παιδιών να μαθαίνουν ξένες γλώσσες και τις ικανότητες των ανθρώπων να βρουν μια θέση εργασίας αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει ένα κύκλο σπουδών σε μια ξένη γλώσσα. Ε, θα σταματήσω γιατί αλλιώς καταχρώμε και το χρόνο σας. Υπάρχουν δυνατότητα να ε, συζητήσουμε περαιτέρω μέσω ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας και ε, γύρω από το θέμα της κοινωνικής ισότητας και τους περιορισμούς στη χρήση της πολυγλωσσίας. Νομίζω ότι αυτές τις στιγμές που ζει η Ευρώπη το θέμα της δημοκρατίας και σε σχέση με την πολυγλωσσία είναι σημαντικό. Ευχαριστώ λοιπόν τους τρεις κύριους ε, ομιλητές εμπειρογνώμονες. Μας έδωσαν μια εικόνα πληρέστατη θα έλεγα Μπορούμε να πούμε σήμερα <clears throat> ότι υπάρχουν συστάσεις, υπάρχουν κάποια μέσα που έχουν ήδη προταθεί εδώ και καιρό. Νομίζω όμως ότι τα ερωτήματα τα οποία παραμένουν είναι πρώτον η συγκρισιμότητα των διαφόρων καταστάσεων στις χώρες που επικρατούν στις διάφορες χώρες μας κάποιες συστάσεις ήδη από το 2008 για την περαιτέρω καθιέρωση της πολυγλωσσίας και σε θεσμικό επίπεδο. Και τέλος, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τους άλλους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που ε, θέτουν μπροστά τους η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να εμβαθυνθούν. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ξεκινήσω με την συνάδελφο Χιμένες από την ομάδα των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συζήτητες για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολυεθνική και πολύγλωση κοινότητα. Έχουμε μια κληρονομιά πολυγλωσσίας, τη φροντίζει και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι κάτι που έχει και οικονομικές επιπτώσεις, αυξάνει την δημιουργικότητα, αυξάνει την καλλιέργεια και επιβεβαιώνει μέσω της πολυγλωσσίας την αξία της διαφορετικότητας. Αυτά τα ακούμε βέβαια και νομίζω ότι και ιδεολογικά μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτές τις, αυτές τις παρατηρήσεις. Βέβαια έχουμε διαφορετικές καταστάσεις στην Ευρώπη. Πολλές φορές οι καταστάσεις οι γλωσσικές οι οποίες υπάρχουν στην Ευρώπη δεν επιτρέπουν την δημιουργικότητα που θα έπρεπε και στην ουσία χρησιμοποιούνται για να δημιουργούν διαφορές και αντιθέσεις στο εσωτερικό των κοινοτήτων. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια πλούσια κληρονομιά, αυτό μας διαφοροποιεί σαν Ευρωπαίους, αυτό είναι και τμήμα της αξίας που έχουμε σαν Ευρωπαίοι, αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λογική αντίληψη γύρω από τις γλώσσες που πολλές φορές δεν είναι εθνικές, δεν είναι μόνο περιφερειακές. Γλώσσες διαπερνούν τα σύνορα και θα πρέπει να δούμε ότι χρησιμοποιούμε επίσης και μια κοινή γλώσσα, μια lingua franca, την οποία προτιμούν μερικές φορές και χρησιμοποιούν οι πολίτες. Η κυρία Φραχάιεν, σας ευχαριστώ και καταρχάς ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει η συζήτηση να διεξαχθεί σε διαφορετικά επίπεδα. Καταρχάς, ε, το τι κάνουμε με την πολυγλωσία στα ίδια θεσμικά μα όργανα και θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον ότι 14 από τις 3 ε, γενικέ διευθύνσει στην Ευρώπη ε, δημοσιεύουν μόνο στα αγγλικά. Δηλαδή, αυτή η πολυγλωσία στην Ευρώπη ουσιαστικά ούτε εμεί θα την προωθούμε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Δεύτερο σημείο. Πώς μπορούμε την πολυγλωσία να την περνάμε και από τα σχολεία, τα διδακτικά συστήματα, από τα συστήματα διαβίου μάθησης, γιατί υπάρχει μεγάλο το του πληθυσμό που είναι μονόγλωσσο. Ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη γλώσσα κατέχει, προκειμένου να μπορεί να διαβάζει, να επικοινωνεί και νομίζω ότι όλη η συζήτηση για το κατά πόσον είμαστε πολύγλωσσοι στην Ευρώπη ή για το κατά πόσον όλοι μιλούν τη γλώσσα τη μητρική τους και έχουν και μία ε, επιπλέον ξένη γλώσσα. Όλα αυτά λοιπόν ε, έχουν να κάνουν και με το εκπαιδευτικό σύστημα σε ό,τι αφορά τα προσόντα και το θέμα ότι δεν συμφωνούμε για αυτά. Αναφέρθηκε επίσης το θέμα του Brexit σε ένα από τα σε μία από τις παρουσιάσεις. Θεωρώ ότι το θέμα του Brexit δεν θα έχει μεγάλη επίδραση σε ό,τι αφορά την αγγλική γλώσσα στην Ευρώπη, γιατί πρόκειται για μία lingua franca. Ακόμα και οι Κινέζοι και στη Λατινική Αμερική ε, μαθαίνει ο κόσμος αγγλικά. Είναι παγκόσμια lingua franca στον επιστημονικό κόσμο, στον κόσμο της τεχνολογία. Είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα γλωσσικά προσόντα και θα πρέπει να κοιτάξουμε και για παράδειγμα το θέμα των γλωσσικών προσόντων ε, των ε, μεταναστών. Για παράδειγμα ε, υπάρχει μια τουρκική κοινότητα αν θέλετε στη Γερμανία η οποία μαθαίνει στα σχολεία γερμανικά και μετά αγγλικά και στα ισπανικά ως ξένη γλώσσα και τελικά δεν μαθαίνει και δεν κατέχει ενδεχομένως καλά τη μητρική του γλώσσα. Άρα και η γλώσσα προέλευσης, η γλώσσα της οικογένειας θα έπρεπε να ενταχθεί πιο πολύ στα σχολικά μας συστήματα. Ο κύριος Μόργανο. Λοιπόν, εγώ καταρχά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τι παρουσιάσει και για την έρευνα που έγινε. Θεωρώ ότι ένα από τα προβλήματα τα οποία θέτει, πρέπει οπωσδήποτε να θέσουμε είναι μια λίγουα φράγκα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω και ως ε, πιο πρακτικές ανάγκες. Και το τι γίνεται σε σχέση με άλλες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη στις Αμερικής. Ένα βασικό του πλεονέκτημα σχετίζεται και με το γεγονό γεγονός ότι έχουμε μια κοινή γλώσσα. Μια σειρά από πράγματα γίνονται βάσει μιας κοινή γλώσσας. Ε, αλλά, όπως είπε και η προναλή σας, θα υπάρξει ένα πρόβλημα αν με το Brexit, ε, όπως έχει ανακοινωθεί, ε, αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορούμε να έχουμε την αγγλική εντό εισαγωγικών ω επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σε πολιτικό επίπεδο δεν θα είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αποφύγουμε, πρέπει να τεθεί. Ε, δεδομένου δε ότι όπως επιθυμήσαμε, Υπάρχει και το γεγονός ότι υπάρχει το θέμα της χρήσης των όρων, ε, νομικά θέματα, οικονομικά θέματα. Επομένως, ε, καταρχήν, σε ευρω... Ε, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο θα τεθεί το ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι η αγγλική δεν είναι γλώσσα από αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται ευρύτατα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι διαφορετική φύσεως το πρόβλημα. Θα είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο ε, κατά πάσα πιθανότητα θα συζητήσουμε ει βάθο. Εκτό μικροφώνου το σχόλιο τη κυρίας Φερχάη. Το πρόβλημα είναι η επίσημη γλώσσα. Γιατί τα Ιρλανδικά... Δεν θα ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση στην παρούσα φάση. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς στο μέλλον θα κληθούμε να συζητήσουμε. Σόιντροβα και μετά ο κύριος Γραμματικάκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν συζητάμε τώρα την πολιτική συζήτηση, δεν κάνουμε την πολιτική συζήτηση της ύπαρξης των Αγγλικών σαν lingua franca, σαν κοινή γλώσσα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Υπάρχουν λοιπόν όπως μας είπαν οι ομιλητές αρκετές μελέτες οι οποίες ε, δείχνουν ποιες είναι οι καλύτερες των πρακτικών τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Δυστυχώς όμως δεν τις ακολουθούμε. Η κατάσταση δεν ε, βελτιώνεται ιδιαίτερα στον τομέα της πολυγλωσσίας. Τα ευρήματα ε, στις συγκεκριμένες έρευνες μας δίνουν ορισμένα στοιχεία αριθμητικά τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Οι στόχοι οι οποίοι έχουν εφητεθεί θα πρέπει να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε νέους κανόνες και νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την πολυγλωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στην παρούσα φάση. Το θέμα είναι να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σημασία για μας είναι η αδυναμία που έχουν ορισμένοι άνθρωποι, η μη δυνατότητα καλύτερα να το πω, να ομιλούν μια κάποια γλώσσα για λόγους πολιτικούς ή κοινωνικούς. Είπατε ότι ένα μεγάλο ποσοστό θα μπορούσαν να επικοινωνούν στα αγγλικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, έναν επιπλέον στόχο σε όλους αυτούς τους οποίους ε, ε, ε, έθεσαν οι εμπειρογνώμονες. Ο καθηγητής Σάβιλ έχετε συχνά εδώ και συμμετέχει στα workshop τα οποία οργανώνουμε και πρέπει να βρούμε ακριβώς τι κίνητρα μπορούμε να δίδουμε και στους νέους και στους μεγαλύτερους σε ηλικία για να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Πρέπει να δούμε πώς τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να ενταθούν μέσα στους προσωπικούς στόχους των νέων, των μαθητών. Αυτά είναι τα πραγματικά μέσα. Πρέπει λοιπόν, καταπολεμώντας και τον αποκλεισμό, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που προέρχονται από μη ευνοημένες κοινωνικές κατηγορίες, που έχουν προβλήματα μεγαλύτερα εκμάθησης, Αυτά τα παιδιά είναι θα έλεγα διατεθειμένα από τη φύση τους καλύτερα να δεχθούν κάποιες προτάσεις. Πρέπει λοιπόν με αποτελεσματικό τρόπο να μπορέσουμε να πείσουμε τις κατηγορίες αυτές τις πιο ευάλωτες να ανοιχτούν σε άλλες γλώσσες όπως και στα αγγλικά. Είπατε ότι ο στόχος μητρική γλώσσα συν 2 είναι ένας καλός στόχος, αλλά πρέπει να υπάρξουν προσαρμογές. Νομίζω ότι αυτός είναι πράγματι ένας στόχος τον οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε. Όμως πρέπει να δούμε ότι το 25% των Ευρωπαίων δεν γνωρίζουν καν καλά τη μητρική τους γλώσσα. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για μας. Δεν θέλω τώρα να φύγω από τη συζήτηση που κάνουμε για ξένες γλώσσες, αλλά όταν μιλάμε για την ποιότητα των μαθημάτων των γλωσσικών, δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι πρέπει να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας και στην διδασκαλία της μητρικής συν μία λίγουα φράγκα ή δυνατόν, συν μία άλλη τρίτη γλώσσα. Είναι μια προϋπόθεση απαραίτητη μεν αλλά όχι επαρκή στο να γνωρίζει κανείς τη μητρική συν μία λίγουα φράγκα, ίσως και μία τρίτη, πολλές φορές ε, είναι κάτι το οποίο δεν αρκεί. Ο κύριος Γραμματικάκης έχει το λόγο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κυρία Πρόεδρε στη σημερινή συνάντηση. Σας συγχαίρω και όσους είχα την πρωτοβουλία. Πρέπει να πω όμως ε, κάποιες παρατηρήσεις. Και οι τρεις εμπειρογνώμονες ήταν πάρα πολύ καλοί παρόλο που καμιά φορά χανόμουν στις λεπτομέρειες. Ε, χανόμουν στη μετάφραση όπως λένε. Ε, ο κύριος Σαβίλ έβαλε το πλαίσιο, ο κύριος Σαβίλ έβαλε το πλαίσιο και το ακολούθησαν. Άκουσα όμως πολύ λίγα πράγματα για κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον για κατά τη γνώμη μου. Και θα παρακαλούσα αν υπάρχει μια απάντηση, ίσως στις παλιότερες εποχές το έχετε συζητήσει. Το πρόβλημα της μετάφρασης σπουδαίων λογοτεχνικών έργων από μικρές χώρες προς γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω πολύ καλά ότι στην πατρίδα μου στην Ελλάδα εφαρμόστηκε ένα τέτοιο πρόγραμμα κατά τρόπο άθλιο και τα βιβλία που μεταφράστηκαν είχαν την τύχη να μεταφραστούν ε, έμειναν στην αφάνεια στην Ευρώπη. Οι γλώσσες όμως οι λογοτεχνικές όπως ξέρετε πολύ καλά και αποδεικνύουν τον πλούτο μιας γλώσσας την κάνουν σεβαστή στις υπόλοιπες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έλεγα μαζί με τη μουσική είναι ένας τρόπος πολύ μεγάλης επικοινωνίας. Δεν ξέρω λοιπόν αν οι αξιότιμοι εισηγητές έχουν κάποια απάντηση σε αυτό. Όπως ξέρετε κυρία Πρόεδρε έχω και προσωπικό ενδιαφέρον διότι έχω γράψει τρία βιβλία για χαριτωμένο το λέω αυτό που είναι όλα bestseller αλλά έχω πολύ δυσκολία να καταλάβω ποιος μπορεί να τα, θα τα μεταφράσει. Ε, Πολύ αυθεντικό αυτό το οποίο είπατε, σημαντικό, γνωρίζετε εν πάση περιπτώσει, ε, ξέρετε, ξέρουμε ότι είστε επιστήμων φυσικός, αλλά ξέρουμε επίσης ότι ασχολείστε και είστε δημιουργικός στον τομέα της λογοτεχνίας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Μαραγάλ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την Ισπανική που δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, τα Καστελιάνο. Δεν είναι ανέκδοτο, γιατί δεν μπορώ εδώ να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Είναι θέμα δικαιωμάτων. Στη δική μου τη γλώτα, γλώσσα και στα, στα Ισπανικά, ε, θα πω ε, σε αυτή τη γλώσσα λοιπόν περίπου αυτό που είπε και η κυρία Χιμένες Μπαρμπάτ προηγουμένως. Η Ευρώπη είναι δημοκρατία και σεβασμό στην ε, ε, ποικιλομορφία. Η κοινή μας γλώσσα, η lingua Φράγκα είναι η δημοκρατία και η lingua Φράγκα μας είναι ο σεβασμός στην ποικιλομορφία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν των πληροφοριών που μας δίνουν σήμερα προώθηση στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, Υπάρχει μια διάσταση που νομίζω ότι δεν εξαντλείται βέβαια σε αυτή τη συνεδρίαση, αλλά είναι παλαχού παρούσα και υπάρχουν και άλλα βήματα και στα οποία θα μπορούσε να συζητηθεί και άλλες ε, εστιάσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε όλα όσα έχουν να κάνουν με τη γλωσσική πραγματικότητα και τη ε, γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Δεν έχουμε την εικόνα του πραγματικού χάρτη της γλωσσικής κατάστασης στην Ευρώπη. Όταν αναφέρεστε σε μητρική γλώσσα, σε τι αναφέρεστε, στις 24 επίσημες γλώσσες ή αναφερόμαστε στις διασταυρώσεις μεταξύ αυτών των επίσημων γλωσσών και των μη επίσημων γλωσσών. Αναφερόμαστε στη σουηδική μειονότητα στη Φιλανδία, στην ουγγρική μειονότητα στην Κροατία, στην Πολωνία ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να είναι. Και αναφερόμαστε στην ποικιλομορφία των ε, λατινογενών γλωσσών. Νομίζω ότι το μόνο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι να έχουμε ένα πραγματικό χάρτη της γλωσσικής ποικιλομορφία. Να έχουμε ένα κατάλογο των γλωσσών και να συσχετίσουμε αυτή την, το χάρτη μητρικών γλωσσών με τα εκπαιδευτικά συστήματα. Η πρώτη απάντηση και η πιο σημαντική είναι να συνδυάσουμε αυτές τις μητρικές γλώσσες με τα ε, αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα και ε, μάλιστα με το μητρική γλώσσα συν δύο ξένες γλώσσες ή συν τρεις ξένες γλώσσες αν θεωρείτε ότι είναι κατάλληλο. Αλλά να ξεκινήσουμε από τη βάση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο ε, σημείο οποιασδήποτε ευρωπαϊκής στρατηγικής από το οποίο δεν μπορούμε να διαφύγουμε. Και υπάρχει και ένα θέμα το είπαμε και ε, προηγουμένως όταν αφαιρθήκαμε σε δικαιώματα, υπάρχουν και θέματα γλωσσικών δικαιωμάτων αναφέρεται και στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται και από την UNESCO ε, στην ορολογία της από άλλη άποψη. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει επαρκής ρύθμιση και δεν έχει εφαρμοστεί επαρκώς ε, ε, το θέμα από τις χώρες μέλη. Το θέμα της lingua franca τα αγγλικά είναι η lingua franca της αγοράς, είναι η lingua franca της οικονομίας και κυρίως της ε, ε, πολιτιστικής κυριαρχίας των Αγγλοσαξώνων στην ψηφιακή ε, εποχή. Δεν προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε κάτι τέτοιο. Είναι εξαιρετικό και αξιοσέβαστο το γεγονός και μακάρι να ήμασταν σε θέση, τουλάχιστον εγώ, να τη χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερη ευχέρεια ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Αλλά νομίζω ότι το θέμα δεν εξαντλείται εδώ, ανεξάρτητα από το αν θα έχουμε Brexit ή όχι. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ε, πολιτικές λύσεις που πρέπει να δοθούν. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η αγγλική είναι αναπόσπαστο τμήμα της συνύπαρξή μας και δεν θα πρέπει ούτε να το λησμονούμε ούτε να το χάσουμε αυτό το μέσο. Επίσης, θα πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την έκθεση Αλφονσή που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 2014 και αναφερθρόταν στο τι σημαίνει πραγματική πολυγλωσία και πώς πρέπει να εφαρμόζεται. Και υπάρχει και μια οικονομική πτυχή και με αυτό ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε. στην ε, αυξανόμενη διάθεση εφαρμοσμένων τεχνολογιών ε, που εφαρμόζονται και στην ε, πολυγλωσία για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη δυνατότητα να μεταφράζουμε, να συμμεριζόμαστε και να έχουμε ανταλλαγή μεταξύ διαφόρων γλωσσών, διότι υπάρχουν αυτά τα εργαλεία δεν είναι μόνο οι εξαιρετικοί διερμηνείς που έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε μέρα έχουμε ε, δίπλα μας μηχανισμούς αυτόματης μετάφρασης, τεχνολογίες που μαθαίνουν. Και επειδή ακριβώς μαθαίνουν είναι και χρήσιμα εργαλεία. Πρέπει λοιπόν να τα χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πράγματι, όταν αναγνωρίζω το πάθος των ομιλητών, προσπαθώ να είμαι γενναιόδοριος προς τον χρόνο, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Τελευταίος ομιλητής και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Τελευταία ομιλήτρια μάλλον. Μποξόρ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Η πολυγλωσία αποτελεί μία μεγάλη αξία στη σημερινή εποχή. Και η πολιτική σε ό,τι αφορά τη γλώσσα θα πρέπει να βασίζεται στην αξία αυτή. Είναι καλή λοιπόν η πρωτοβουλία ότι ακολουθούμε αυτή την αρχή της μητρικής γλώσσας σε δύο α, ξένες γλώσσες. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άτομα που ζουν και είναι σε ομάδες Δηλαδή έχουν τη μητρική τους ε, γλώσσες, ε, συνδύο ξένες γλώσσες, αλλά πρέπει να μάθουν και τη μητρική γλώσσα, τη γλώσσα του κράτους τους δηλαδή. Και τελικά καταλήγουμε σε τουλάχιστον τέσσερις γλώσσες. Αυτό έχει να κάνει και σε σχέση με αυτά, έχει να κάνει και με αυτά που είπατε προηγουμένως, κύριε Φερχάιρν, για την τουρκική κοινότητα, για παράδειγμα. Και ο κύριος Μαραγκάλα ανέφερε παραδείγματα σχετικά. Αυτό θεωρώ ότι ισχύει και για τους Ουγγρούς στη Ρουμανία, στη Σλοβακία, στην, ε, σε, άλλες γλώσσες, σε άλλες χώρες όπου αποτελούν γλωσσική μειονότητα. Και θα χρειαζόντουσαν θεωρητικά ε, έρευνες, μελέτες για να διαπιστώσουμε σε τι κατάσταση γλωσσική βρίσκονται οι μειονότητε αυτέ και τι δυνατότητε έχουν να μάθουν τι γλώσσε κτλ. Αλλά δεν ε, έχει ανακοινωθεί η διεξαγωγή τέτοιων συγκεκριμένων ερευνών. Θα ήταν καλό να υπάρχουν όμω οι έρευνε αυτέ με συγκεκριμένα πορίσματα τα οποία θα λαμβάναμε υπόψη. Πέρα από τα αγγλικά επίση, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η πιο δημοφιλή γλώσσα. Υπάρχουν στοιχεία προ την κατεύθυνση αυτή. Ε, από ό,τι βλέπετε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον μετά τι παρουσιάσει σα, και το θέμα αυτό είναι ανοιχτό. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα ε, πολλών ζητάσεων, υπάρχει εφαρμογή, επαληθεύουμε κατά πόσον τα κράτη-μέλη ε, υιοθετούν πράγματι όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν νέε προκλήσεις λοιπόν και βλέπουμε και τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας. Και πιστεύω, και εδώ θα είναι πελίτημο να ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι στην πραγματικότητα εσείς ξανανοίξατε τις διάφορες εκδοχές. Όταν αναφερθήκατε στις τρεις προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει, όταν εσείς είπατε πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει συνέπεια μεταξύ κινητικότητας και κοινωνικής ένταξης ε, μέσω της γλωσσικής ποικιλομορφίας και όταν αναφέρετε και ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα εργαλεία εκμάθησης γλωσσών. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ προκειμένου να μπορέσουμε να ακούσουμε και τη δική του την άποψη για τη συζήτηση και ο λόγος είναι στην κυρία, συγγνώμη θα το βρω το όνομά σας, Σοφή Μπερνάρ, σε τμήμα, τμήματάρχη της Γενικής Διεύθυνσης και μετά ο Λούκα Τομάζε. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είμαι από τη Γενική Διεύθυνση που ασχολείται με θέματα σχολείων και πολυγλωσίας να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που παρουσίασαν ένα εξαιρετικό πανόραμα των πρωτοβουλειών που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογράμμισαν αυτά τα οποία μπορέσαμε να πετύχουμε σε επίπεδο πολιτικής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, όπως επίσης και τις έρευνες οι οποίες έγιναν τα τελευταία χρόνια. Δεν θα επανέλθω σε αυτά, το έκαναν καλύτερα. Άκουσα επίσης ε, πολλές συστάσεις, τρεις τύπους θα έλεγα συστάσεων. Πρώτος, είναι η συνέχιση της πολιτικής συνεργασίας στον τομέα της πολυγλωσσίας, συνέχιση της δουλειάς την οποία κάνουμε, λαμβάνοντας υπόψη το λεγόμενο νέο περιβάλλον. Υπογραμμίσατε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, την κινητικότητα, και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Συνεργαζόμεθα με εμπειρογνώμονες σε σχέση με τις λεγόμενες πολύγλωσσες τάξεις και την δυσκολία που υπάρχει στις τάξεις αυτές όπου διδάσκεται η γλώσσα διδασκαλίας και ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η, η γλώσσα προέλευσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές από τις διάφορες χώρες. Υπογραμμίσατε στην αρχή της συνάντησης τα συμπεράσματα στα οποία είχαμε καταλήξει την Ευρωπαϊκή ημέρα των γλωσσών τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Πράγματι εκεί δόθησαν ορισμένοι προσανατολισμοί οι οποίοι δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των λεγόμενων peer learning activities, δηλαδή συνεργασία με εμπειρογνώμονες των Υπουργείων Παιδείας. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να δούμε σε ποιο βαθμό τα προγράμματά μας έχουν αποτελέσματα και σε ποιο βαθμό μπορούν να μεταφερθούν επίσης ε, ε, και σε άλλες χώρες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, είναι κάτι το οποίο αξιολογείται συστηματικά πριν καταλήξουμε σε προγράμματα τα οποία ε, θα έλεγα συγκεντρώνουν την προτίμησή μας. θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτές οι σημάνσεις πολλές φορές δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς διευρύνουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και καταλήγουμε σε πολιτικά συμπεράσματα ενδιαφέροντα, αλλά λειτουργούμε κυρίως σε επίπεδο διάδοσης. Συνεπώς χρηματοδοτούμε και έρευνες όπως αυτές τις οποίες αναφερθήκατε από το ΚΡΕΛ, ή από ε, συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης για να κρίνουμε σε ποιο βαθμό η εκμάθηση ξένων γλωσσών επηρεάζει την απασχολησιμότητα. Συνεχίζεται η προσπάθεια, θεωρούμε ότι είναι ο τομέας αυτός πολλά υποσχόμενος. Ένα τρίτο θέμα που υπογραμμίστηκε είναι ανάγκη περαιτέρω διάδοσης, καλύτερης κυκλοφορίας των μελετών στον κόσμο. Αυτό γίνεται, δεν είναι αλήθεια ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Διαδίδονται τα προγράμματά μας, θα πρέπει να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω στα προγράμματα αυτά για να καθορίσουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη κάποιες πολιτικές οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έγιναν επίσης πολλές συζητήσεις σήμερα για το lingua franca, αγγλικά ή όχι κτλ. Αυτό το οποίο θα έλεγα υπογραμμίστηκε και σωστό ήταν, είναι το πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνει κανείς τις γλώσσες ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο ζει. Κάποιος ο οποίος ζει σε μια μεθοριακή περιοχή προφανώς έχει ενδιαφέρον να μάθει τη διπλανή γλώσσα παρά τα αγγλικά αυτό επηρεάζει άμεσα άλλωστε τη δυνατότητα συμμετοχής ε, στις, στην αγορά εργασίας στις δύο χώρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει η κυρία Κώστα. Δύο σκέψεις και θα δώσω το λόγο στους ομιλητές για να κλείσουν τη συζήτηση. Πρώτον, όπως ε, προτείνατε κι εσείς, αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι οι πολιτικές τις οποίες ακολουθήσαμε μέχρι τώρα και θα πρέπει ε, να ενταχθούν στην λεγόμενη ε, skill agenda, δηλαδή ποιες είναι οι στρατηγικές και πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις γνώσεις και τις δυνατότητες των εργαζομένων. Αυτά είναι θέματα που άπτονται και των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτισμού. Βλέπω επίσης ότι τον, στις επιμέρους γλώσσες υπάρχει μια ένδια σταδιακά σε σχέση με τις περιφερειακές και τις λιγότερο μιλούμενες γλώσσες. Και μια παρατήρηση το έθεσε ο κύριος Γραμματικάκης, είναι και το θέμα της λογοτεχνίας, είναι το θέμα της διάδοσης, δηλαδή των πολιτισμών μέσω των γλωσσών. Η γλώσσα της μετάφρασης δηλαδή δεν είναι μόνο μία γλώσσα, αλλά είναι και κάτι το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλους πολιτισμούς και πρέπει να ευνοηθεί. Και υπάρχουν επίσης και κάποιες γλώσσες οι οποίες για λειτουργικούς λόγους μελετώνται περισσότερο, αγγλικά ίσως. Ε, η δική μου γλώσσα, η ιταλική γλώσσα, είναι η τέταρτη υποτίθεται που μελατάτε στον ε, κόσμο. Όχι ότι είναι και πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά για λόγους πολιτιστικούς, ιστορικούς. Ε, για λόγους θα έλεγα που βασίζονται σε συναισθήματα απέναντι σε μια κουλτούρα, σε μια χώρα, σε μια ιστορία. Λοιπόν, αυτό αυτά. Βλέπουμε ότι η γλώσσα και ο πολιτισμός πηγαίνουν μαζί. Θα σεβαστώ τη σειρά με την οποία μιλήσατε προηγουμένως. Ο κύριος Σάβιλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που προσπαθούμε να καλύψουμε πάρα πολύ ε, έδαφος, πάρα πολύ μεγάλη ύλη σήμερα το πρωί και εγώ θα σας έλεγα να κοιτάξετε τις μελέτες γιατί υπάρχουν πολλές ε, πληροφορίες τις οποίες δεν σας αναφέραμε, δεν προλάβαμε και αυτές απαντούν ε, σε κάποιο βαθμό τις ερωτήσεις σας, ε, τα σχόλια που κάνατε και μεταξύ άλλων και τη δουλειά που κάναμε στα πλαίσια των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν να κάνουν με τη μετάφραση. Και κάτι που θα ήθελα να τονίσω στα συμπεράσματά μου, στα απορίσματα μου εγώ έδειχνα ε, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ο κόσμος, ε, όπου θα σκεφτόμασταν αυτό το μητρική γλώσσα συν δύο ξένες γλώσσες, γιατί είναι μάλλον απλοϊκή, αν θέλετε, αντίληψη της γλωσσικής ε, πολυμορφίας αυτό. Είναι ένα σαφή στόχο, βέβαια, αλλά προφανώ ε, ε, εμπλέκονται και πολλά ζητήματα. Όπω αυτά που αναφέρατε. Τι σημαίνει μητρική γλώσσα, ποια είναι η γλώσσα του σπιτιού, ποια είναι η γλώσσα τη εκπαίδευση και τι γλώσσα θέλει να μάθει κανεί ω άτομο ε, στη ζωή του. Για να έχει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες επικοινωνίας. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει το να μαθαίνει κανείς γλώσσες, για παράδειγμα, για πολιτιστικούς σκοπούς ή για άλλους λόγους. Και αυτό καθορίζει τελικά τη γλωσσική ταυτότητα του καθενός. Κάτι προσωπικό, όχι κάτι το οποίο στο βάζει κανείς ως ετικέτα. γαλλόφωνο, ταλόφωνος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με την προσωπική πολυγλωσία. Αυτό που αναφέρεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως plurilingualism, πολυγλωσία. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές ικανότητες και στι διαφορετικές γλώσσες. Δεν είναι πλήρης οι ικανότητες σε όλες τις γλώσσες. Χρειάζεται κανείς μια γλώσσα για κάποιους σκοπούς. Για παράδειγμα το να μιλάει κανείς τη γλώσσα του σπιτιού, να μιλάει τη γλώσσα των γονιών, των παππούδων, να μιλάει κανείς τη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, να ταξιδεύει, να υπάρχει μια lingua franca που θα τον βοηθάει να επικοινωνεί σε άλλες χώρες και μετά στην ε, ε, εργασία, ενδεχομένως να υπάρχει μια νέα γλώσσα. Δεν υπάρχει ένας προδιαγραμμένος δρόμος προς τα εμπρός. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμπνεύσουμε τους νέους ανθρώπους να μάθουν γλώσσες. Και αυτό είναι η αποτυχία, αν θέλετε, του σχολικού συστήματο. Το να βάλουμε τα παιδιά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να του λέμε μάθε αυτή τη γλώσσα δεν ωφελεί ιδιαίτερα. Θα πρέπει να βγουν πέρα από τα τετριμένα και να δουν τι γλώσσε ω κάτι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι, στην κοινωνία, στην ε, αγορά εργασία. Ε, νομίζω ότι με πολλού τρόπου μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά σίγουρα η τεχνολογία θα μα βοηθήσει ιδιαίτερα. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο προλαλής σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν συζητούμε πολιτική, ε, γλωσσική παιδεία και με την ευρία έννοια, Αναφερόμαστε συχνά στις γλώσσες και σπανίως στους ανθρώπους. Κατά την άποψή μου, όσο περισσότερο αναφερόμαστε στους ανθρώπους και στις δυνατότητες ε, να αναπτύξουν ε, τις γλωσσικές τους δεξιότητες, που πάντα είναι ε, επαρκής, καλό είναι να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες λύσεις, αλλά και τοπικές. Οι τοπικές λύσεις είναι οι καλύτερες. Επομένως, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφός μου. Πρέπει να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα άτομα και να υποστηρίζουμε την γλωσσική τους ανάπτυξη, να τους ενθαρρύνουμε να αναπτύξουν τις δυνατότητες που έχουν γενός στα γλωσσικά, κατά τρόπον ώστε να συμμορφώνονται περισσότερο στις προσωπικές και κοινωνικές τους ε, ε, καταστάσεις και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζουν. Ακόμα και από τον υπηαγωγείο μέχρι τη θέση εργασίας θα πρέπει να γίνεται αυτό. Όταν θα πρέπει ε, πλέον το άτομο να δρά προς όφελος της κοινωνίας. Πάρα πολύ σύντομα πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διάκριση ανάμεσα στα όργανα τα ευρωπαϊκά, αυτό που πρέπει να κάνουν και τις ανάγκες των πολιτών σε επίπεδο προσωπικό και επαγγελματικό. Τα ευρωπαϊκά όργανα χρησιμοποιούν σαν πρότυπο και τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά κυρίως πρέπει να δουν τι γίνεται σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Ελβετία, με ε, σωστή διαχείριση της πολυγνωσίας, τη απουσία μιας λίγκουα φράγκα, ε, όπου τα τοπικά όργανα και οι κυβερνήσεις γνωρίζουν τι θέλουν οι πολίτες τους. Πρέπει να δούμε τι έχουν ανάγκη οι πολίτες στην ζωή τους σε επίπεδο γλωσσικό. Η Ευρώπη δεν είναι μια ελληνικού τύπου, αρχαιοελληνικού τύπου αγορά είναι ένα περιβάλλον στο οποίο ναι μεν οι πολίτες μετακινούνται ελεύθερα, αλλά οι γλωσσικές ανάγκες αλλάζουν. Να σας δώσω ένα πλαίσιο για να καταλαβαίνετε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Ο Υπουργός Παιδείας της Ολλανδίας είπε πρόσφατα ότι μόνο το 30% των ξένων φοιτητών που σπουδάζουν στην Ολλανδία στα αγγλικά μένουν εκεί για να εργαστούν, μόνο το 30% ενώ θα ήθελαν το 70% να το κάνουν και αυτό οφείλεται στις γλωσσικές ελλείψεις που έχουν στην Ολλανδική γλώσσα. Συνεπώς βλέπετε ότι υπάρχει μια περιπλοκότητα στον τομέα των γλωσσικών, η οποία δεν πρέπει να ερμηνεύεται με απλοποιημένο τρόπο. Θα πρέπει να δούμε ε, τι υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε ε, για παροχές εννοώ σε επίπεδο γλωσσικές σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και όχι σε σχέση με αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς χρήσιμο. Για την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει μεγάλη σημασία να μην ζητήσουμε μόνο από αυτούς που χρηματοδοτούν ε, τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά να προβλέψουν το τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό το οποίο ήθελα να πω εγώ είναι να υπολογίσουμε λίγο τα αποτελέσματα εκ των υστέρων. Τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των γνώσεων των ανέργων. Έδωσε αποτελέσματα, ωφέλησε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα πλατφόρμα, αλλά θέλουμε να συγκρίνουμε τις πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται και στον τομέα των γλωσσικών πολιτικών. Ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις σας, ανοίξατε περαιτέρω σενάριοι Γίνεται επίσης και μία έρευνα σε αυτή τη φάση για τις γλωσσικές μειονότητες. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες και εκεί. Πρέπει να ορίσουμε ακριβώς ε, σε τι ε, αναφερόμαστε. Αναφέρθηκε ε, σε αυτά και η κυρία Μπόξορ και άλλοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε όλους. Νομίζω ότι στα πλαίσια των ικανοτήτων των εργαζομένων θα πρέπει ίσως να χρησιμοποιήσουμε και τις δικές σας προτάσεις. Δεν θέλουμε να χάσουμε την εμπειρογνωμοσύνη σας με κανένα τρόπο. Η συνάντηση νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ. Take the seat Είναι η τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς και όλοι είναι λίγο αναστατωμένοι. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Νομίζω ότι έχετε όλοι ενδιαφέρον να συζητήσετε τα θέματα που έχουμε μπροστά μας. Ε, eh, eh, λοιπόν, ξεκινάει η πρώτη συζήτηση για το Creative Europe. Είμαι εισηγήτρια γι' αυτό. Θα ήθελα σαν πρόεδρος πάντα να πω ότι ευχαριστώ για την παρουσία τους, για την Digit Connect, τον κύριο Τόζον, αναπληρωτή ε, τμήματάρχη, ο Καρελ Μπάρκ είναι ο υπεύθυνο και τον κύριο Σιμάνοβιτς, πάντα από την DG Connect και από την ΕΣΕΑ είναι ο Brian Holmes, διευθυντής. Τον συναντήσαμε πρόσφατα όταν επισκεφθήκαμε την ΕΣΕΑ με την αρμόδια επίτροπο. Μετά τη δική μου παρέμβαση θα δώσω το λόγο στη Γενική Διεύθυνση για να μας δείξει τα καινοτόμα στοιχεία μετά τη συμφωνία της DG Connect και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ε, νομίζω ότι Μέχρι τον Ιούνιο, τέλος του μηνός, θα υπάρξει συμφωνία. Έχουν διανεμηθεί τα έγγραφα. Θα δώσω πρώτα το λόγο, μετά την παρέμβασή μου δηλαδή, στους δύο προσκεκριμένους. Μετά θα μιλήσουν οι σκιώδεις και μετά εκ νέου τον λόγο στην Επιτροπή. Το Creative Europe εφαρμόστηκε ήδη από τον Ιανουάριο του 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τον επόμενο χρόνο τα ενδιάμεσα αποτελέσματα. Αλλά όπως ξέρετε εμείς για πρώτη φορά θα έχουμε το Erasmus Plus και για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο αποφάσισε να έχει ε, εκθέσεις ε, που θα εξετάζουν την εκτέλεση των προγραμμάτων και επιτρέπουν και σε εμά ως εισηγητές ε, να μπορέσουμε ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, αλλά και να έρθουμε και σε επαφή με ενδιαφερομένους και ισχυώδεις εισηγητές, να μιλήσουμε και με τις εθνικές υπηρεσίες και φυσικά και με όλους τους διαφόρους συνομιλητές προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε και γέρος και κάποιες κατευθύνσεις, ε, να επαληθεύσουμε κατά πόσον εφαρμόστηκε σωστά το πρόγραμμα και κάποιες ε, συστάσεις για το μέλλον. Βάσει προγράμματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Ε, στην επόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση θα πρέπει να εξετάσει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ε, προγράμματος και την επίτευξη των στόχων, την αποδοτικότητά του και σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, να περιλαμβάνει ε, και την αξιολόγηση του κόστους, την προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, ε, η απλούστευση που τη χρησιμοποιούμε συνέχεια αλλά ποτέ δεν υλοποιείται, την εσωτερική συνοχή του προγράμματος, το κατά πόσον είναι είναι σχετική ακόμα η στόχη, το κατά πόσον συνεισέφερε το πρόγραμμα στην επίτευξη των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για μια ευφυή ε, βιώσιμη και ε, ανάπτυξη που περιλαμβάνει τους πάντες. Η έκθεση λοιπόν για την, ε, ο Κοινοβούλιο που θα σας παρουσιάσω θα πρέπει να δει κατά πόσον το πρόγραμμα ακολουθεί τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό και πώς εφαρμόζεται στη δεύτερο τμήμα της έκθεσης θα πρέπει ε, να ε, φανεί και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και σε μια περαιτέρω συζήτηση, όχι μόνο σήμερα, για να σας πω και λίγο τι θα κάνουμε στη συνέχεια, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να ξανασκεφτούμε ίσως το πρόγραμμα για να το προσαρμόσουμε στις νέες απαιτήσει και να θέσουμε τις βάσεις για την επόμενη επταετία, ίσως και με διαφορετικό τρόπο. Ε, με τη γραμματεία ε, ζητήσαμε τρεις μελέτες, ε, δύο από τις οποίες έγιναν από το Τμήμα Πολιτικής και αφορούν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο υπευλήθη στα Εθνικά Γραφεία της Δημιουργικής Ευρώπης που αφαιρούσε το ένα το υποπρόγραμμα ε, για τον πολιτισμό και το άλλο το υποπρόγραμμα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η τρίτη μελέτη έγινε από την ε, ε, Υπηρεσία Τεκμηρίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι διαθέσιμο για όλους τους συναδέλφους, το έχουμε και εδώ στην αίθουσα. Αποφασίσαμε σήμερα... Ε, να κάνουμε και μία ε, συζήτηση και να παρουσιαστούν όμως και τρεις μελέτες για να έχουμε όλα τα στοιχεία, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου, γιατί θα είναι και πιο εύκολο φυσικά, ε, ε, θα έχουμε και παρουσία συναδέλφων που σήμερα δεν μπορούσαν να παρευρεθούν, θα παρουσιάσουμε λοιπόν τις μελέτες και θα εμβαθύνουμε και σε αυτά. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω κάποιες δικές μου σκέψεις και κάποιες παρατηρήσεις μετά από μια σημαντική συζήτηση και διαβούλευση που κάναμε. Μιλούσαμε με αρκετού ενδιαφερομένους, ε, συναντήσαμε ενδιαφερομένους ε, του, των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού, του συντονιστές των εθνικών γραφείων ε, και κάποιους εθνικούς φορείς στον τομέα του πολιτισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της δημιουργικής βιομηχανίας, καθώς επίσης και μια συνάντηση που θα κάνω τον Οκτώβριο στη Γαλλία ε, για να ακούσω και λίγο και την πραγματικότητα για το πώς ε, εκτελέστηκε το πρόγραμμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Δημιουργική Ευρώπη ενωπεί τρία προγράμματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη επταετία, ε, κουλτούρα, μέντια και μέντια μούντους, όλα αυτά συνενώθηκαν με κοινούς στόχους που διαρθρώνονται όμως και έχουμε δύο υποπρογράμματα και δύο διατομιακά στοιχεία. Έχουμε συγκεκριμένους στόχους και πολύ συγκεκριμένο και προπολογισμό και ποσόστοση για το καθένα καθένα. Έτσι μπορέσαμε να έχουμε στοιχεία σύγκληση μεταξύ του πολιτιστικού, του δημιουργικού και του οπτικοακουστικού τομέα και βεβαίως ε, βλέπουμε και πώ συνεισφέρουν στην ε, ανάπτυξη και στην ε, κοινωνική ένταξη. Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνεται και από τα οικονομικά στοιχεία του τομέα Έχουμε συνεχή ανάπτυξη, πολύ πάνω από τους γενικούς στόχους και μάλιστα η έκθεση η οποία παρουσιάστηκε για τη δημιουργική βιομηχανία στη συζήτηση που έγινε μεταξύ πολιτισμού και ε, Ήτρε αναφερθήκα σε 12.000 θέσεις εργασίας ε, ευρύτερα από τους κλάδους αυτούς που είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Θεωρήσαμε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει μια εγκάρσια διάσταση του πολιτισμού που είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Τι συνέβη. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα δομή της Επιτροπής Juncker ανέθεσε τη διαχείριση τη Δημιουργική Ευρώπη σε δύο διαφορετικού επιτρόπους και σε δύο διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει: την ΕΑΚ και την CONNECT. Και παρά το γεγονό ότι σε κάποια πράγματα υπάρχει πολύ μεγάλη δέσμευση για κοινή εργασία, υπάρχει και μια διαφοροποίηση στην προσέγγιση και ορισμένε δυσκολίε ε, προκειμένου να υπάρχει μια κοινή ε, κατεύθυνση και κάποια κοινά κριτήρια και ε, λόγω και τη φυσική τάση του Μέντια να επενδύει κυρίω στην ε, οπτικοακουστική βιομηχανία και το πρόγραμμα του Σκουλτούρα για να επενδύσει στον τομέα των μη κυβερνοσκοπικών ε, οργανώσεων και στη νέα δημιουργική βιομηχανία. Ο τομέα όμω των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών, που δεν είναι οπτικοακουστικέ, μουσική, εκδόσει, αρχιτεκτονική, σχεδιασμό, ε, βιοτεχνία, για να αναφερθώ σε κάποια, δεν εκπροσωπούνται επαρκώ στο Κουλτούρα και θα χρειαζόντουσαν περισσότερη συγκεκριμένη προσοχή. Εδώ έχετε να προσταθεί και το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε η ε, διακλαδική διαδικασία που είχαμε σκεφτεί για να υποστηρίξουμε ολοκληρωμένα και καινοτόμα προγράμματα. Και ξέρουμε ε, ότι υπάρχουν περιορισμένοι πόροι μεν, αλλά πρέπει να το πούμε. Χρησιμοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά για να υποστηρίξει το πρόγραμμα. Τα γραφεία, την έρευνα, την επικοινωνία κλπ. Επίσης, να πω και τα υπόλοιπα τώρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η καστηθέρηση για το ε, μέσο εγγύηση για τις δανειοδοτήσεις που έχει 30, 120 ε, εκατομμύρια ευρώ για να επενδύσει στα επόμενα 6 χρόνια. Ελπίζω να γίνει επιλογή μέχρι τον Ιούλιο για να υπάρξουν μειοδοτικοί διαγωνισμοί και να υπάρξουν ε, ε, και κατάλληλα ε, θέματα τα οποία θα υποβληθούν και θα είναι προσαρμοσμένα στη δημιουργική βιομηχανία και στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και να υπάρχει και ένας άλλος μειοδοτικός διαγωνισμός για να βρούμε ποιος ε, ε, θα υποστηρίξει τις δυνατότητες ε, των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρωμάτων για να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες του τομέα. Η καθυστέρηση φυσικά σημαίνει ότι δεν έχουμε στοιχεία για να δούμε κατά πόσον αυτή η καινοτομία του προγράμματος είχε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Δεν τα είχε ήδη γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Έχουμε κάποιες δυσκολίες, έχουμε καθυστέρηση και θα καθυστερήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου να μας πει τα αποτελέσματα. Ελπίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή διαχείριση που θα ε, είναι συνδυασμένη μεταξύ των Γείων Γενικών Διευθύνσεων θα μα βοηθήσουν να έχουμε μια αποτελεσματική συνεργασία και να έχουμε και αυτή την ισορροπία που ζητάμε μεταξύ του μη κερδοσκοπικού και του κερδοσκοπικού τομέα. Η ε, Δημιουργική Ευρώπη για την επταετία 2014-2020 στον τίτλο 3 του ε, προγράμματος πλαίσιο είναι 1,46 εκατομμύρια ευρώ και είναι το 0,14% του συνολικού προπολογισμού του πολέτου δημοσιονομικού προγράμματο. Από τη συνολική προοικοδότηση, το 31% διατίθεται στο υποπρόγραμμα Κουλτούρα, το 56% στο Μέντια και το 13% στο ε, διακλαδικό σκέλος. Πρέπει να πω ότι οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί, μετά από κάποιες έρευνες, ε, έχουμε και τα σχετικά στοιχεία, ε, ξεκίνησαν εγκαίρως παρά το γεγονός ότι αρχικώς είχαμε μια καθυστέρηση και έχουμε ε, ε, περίπου 100% του προϋπολογισμού και για τις δεσμεύσεις αλλά και για τις πληρωμές. Ε, ε, για το προϋπολογισμό του 2017 έχουμε μια μικρή αύξηση, είμαστε στα 201 εκατομμύρια και το γνωρίζουμε ότι δεν αρκούν αυτά τα κονδύλια για να μπορέσουμε να έχουμε την ανάπτυξη που ε, μπορεί να επιφέρει η Δημιουργική Ευρώπη. Αυτή είναι πολιτική δήλωση και με τους συναδέλφους χθες τα συζητήσαμε τα πράγματα αυτά. Από το 14 στο 2015 χρηματοδοτήσαμε 351 προγράμματα ανάμεσα σε 1.691 προτάσεις, δηλαδή 20% του ποσοστού. Έχουμε ένα ποσοστό το οποίο εγώ βρίσκω 11% ε, αποδοχής, άλλοι θεωρούν 13% για το κύριο πρόγραμμα, το πρόγραμμα συνεργασίας και 6% για την πλατφόρμα. Για το Μέντια, το οποίο χρησιμοποιεί άλλα κριτήρια σε σχέση με το τομέα της διανομής, σαν παράδειγμα, χρηματοδότησε 4.494 προγράμματα μετά από 8.471 αιτήσει, δηλαδή 43%, πολύ ψηλό ποσοστό κάλυψης. Αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί διαφορετικά λοιπόν σε αυτούς που ασχολούνται με τα προγράμματα αυτά. Είναι στην ουσία θύμα της επιτυχίας τους. Πολλές φορές αποκλείονται προγράμματα για 0,5 βαθμού. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί, αν θέλετε, μια μορφή άρνηση σε σχέση με την κατάθεση των προγραμμάτων ε, στα πλαίσια των προϋπολογισμών του 2017 θα ολοκληρωθούν με καλύτερο τρόπο οι διαθέσιμες πιστώσεις. Τώρα από όλε τις συναντήσεις τις οποίες κάναμε μέχρι τώρα τι μπορούμε να δούμε, τι μπορούμε να βρούμε. Συναντηθήκαμε με τους επιτρόπους, με την EAC, ε, ε, ε, με το DESK κτλ. Ευχαριστώ για τον διάλογο και την διαθεσιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πήρα μέρος επίσης στο Cultural Fund των Βρυξελών, του Βερολίνου, στο Film Forum του Βερολίνου και επισκέφθηκα και διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πήρα μέρος και στην απονομή των βραβείων για τις ετικέτες, για την κληρονομιά και για την λογοτεχνία θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω κάποια επιμέρους στοιχεία. Θα έλεγα το οικονομικό κομμάτι και το κομμάτι του marketing είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί εις βάρος του περιεχομένου, της ποιότητας και της καινοτομίας. Αυτή είναι η αντίληψη την οποία έχουν όσοι συμμετέχουν. Θα πρέπει εμείς να μην υποκύψουμε σε παλαιού τύπου οικονομικίστικες λογικές και θα πρέπει να λειτουργήσουμε με, ε, εφάνταστο και ε, δημιουργικό τρόπο. Οι δείκτες οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί από την Γενική Διεύθυνση ΕΑΚ δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικοί και προβλέπονται πολλές φορές μέσω των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό δημιουργεί κινδύνους για το μέλλον του προγράμματος γιατί δεν θα είναι σε θέση να υπογραμμίσει τις δυνατότητες που έχει. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της καθυστέρησης του χρηματοδοτικού μέσου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να κλείσει το μέσο ε, του Media Mundus λέγοντας ότι το πρόγραμμα αυτό θα είναι ανοιχτό σε όλες τις χώρες και σε τρίτες χώρες μέσω διμερών συμφωνιών. Είναι σαφές όμως ότι σε σχέση με αυτό θα πρέπει να γίνει μια θα έλεγα προσπάθεια διάδοσης, γνωστοποίησης, διαφήμισης γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να υπάρξει ενδιαφέρον και σύν της άλλης θα είναι και γεωγραφικά α, μη ισορροπημένο. Δεν υπάρχει ούτε ένα πρόγραμμα από χώρες του Νότου, ε, ενώ του Νότου της Μεσογείου. Υπάρχουν χώρες όπως η Γεωργία, η Ουκρανία, η Σερβία, αλλά απαιτείται να υπάρξουν και άλλες ε, προελεύσεις θα έλεγα ενδιαφέροντος. Το υποπρόγραμμα για τον πολιτισμό λοιπόν και αυτό θέτει ορισμένους προβληματισμούς. Είναι ενδιαφέρον πρόγραμμα, συνεισφέρει στην κοινοτικότητα των καλλιτεχνών, δημιουργών κτλ. Καταρχάς υπάρχουν τα δίκτυα τα οποία έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο αλλά έχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με την επιλεκτικότητα. Η νομική του φύσης, η παλαιότητα ε, και άλλες τεχνικές λειτουργίες δημιουργούν προβλήματα. Οι πλατφόρμες ε, είναι πολλά υποσχόμενες αλλά έχουν μικρό μέγεθος. Οι λογοτεχνικές μεταφράσεις πρέπει να τύχουν ενίσχυσης από εδώ και πέρα και μέσω του Ευρωπαϊκού Βραβείου για την Λογοτεχνία και σε συνεργασία με τις εκδοτικές δραστηριότητες και όχι μόνο για τις μικρές γλώσσες αλλά και για τις μεγαλύτερες. Στον τομέα της συνεργασίας υπάρχει μια κάποια μορφή ολοκλήρωσης ανάμεσα στους τομείς, ιδιαίτερα σε τομείς όπου κυριαρχούν ορισμένες δραστηριότητες όπως ο τηλεοπτικός κτλ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον να προσπαθήσει κανείς να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, να προσπαθήσουμε να δούμε δηλαδή ένα νέο υποπρόγραμμα για τις δημιουργικές και καλλιτεχνικές βιομηχανίες, μουσική, design, ε, καλλιτεχνική δημιουργία, καλλιτεχνική βιοτεχνία και να αφήσουμε το θέμα της συνεργασίας στα πραγματικά νομικά αν θέλετε πρόσωπα. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στο μέλλον για μετά το 2017. Τώρα για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του πολιτισμού. Ο νέος κανονισμός από το 2014 ε, δείχνει τρεις τέτοιες πόλεις τον χρόνο. Έχουμε επίσης ε, και την ευρωπαϊκή ετικέτα αν θέλετε και τα ευρωπαϊκά βραβεία για την αρχιτεκτονική, την κληρονομιά, την λογοτεχνία. Έχουμε επίσης και το Border Breakers και πρέπει να ξανά έλθει το βραβείο για το θέατρο. Έχουμε επίσης για τον κινηματογράφο και το βραβείο Λούξο για το Μέντια το Μέντια εξακολουθεί να υποστηρίζει τον ε, ραδιοτηλεοπτικό και οπτικοακουστικό γενικότερα τομέα, παρέχει προστιθέμενη αξία, δημιουργεί μάλλον προστιθέμενη αξία. Στο τελευταίο φεστιβάλ στις Κάνες 23 έργα υποστηρίχθηκαν από το Μέντια και 11 από αυτά βραβεύθηκαν. Τα παιδιά του Σαούλ, βραβείο Όσκαρ του 2016, χρηματοδοτήθηκε από το Μέντια. Αυξήθηκαν επίσης και τα εισιτήρια που έκοψαν οι ταινίε αυτές, έφτασαν τα 980 εκατομμύρια και το 30% είναι ευρωπαϊκά κινηματογραφικά έργα. Συνεπώς αυτό επηρεάζει τους παραγωγούς. Τα 12 αν θέλετε τμήματα του Μέντια είναι πολύ γνωστά και καλοδεχούμενα στον δημιουργικό τομέα θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια για το θέμα το λεγόμενο της audience development, της ανάπτυξης του ακροατηρίου. Υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να ειδωθούν και στον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και σε σχέση με τον οποίο βαθμολογούνται αν θέλετε σε κάποιες ισχυρές χώρες στον τομέα της παραγωγής κινηματογράφου για να βοηθηθούν οι ασθενέστερες χώρες. Αυτά τα χάντικα που ουσιαστικά είναι ε, ιδιαίτερα υψηλά για κάποιες χώρες και δημιουργούν στρεβλώσεις θα έλεγα για χώρες οι οποίες ε, έχουν δυνατότητες εξαγωγικές στον κινηματογράφο τους και δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Τώρα στον διακλαδικό ή διατομεακό χώρο αν θέλετε Υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι τα μεμονωμένα προγράμματα, τα διατομεακά ή διακλαδικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε και υπό το φως του εισαγόμενου, θα έλεγα, πολιτισμού για από πλευρά των μεταναστών, των πολιτιστικών στοιχείων, θα πρέπει ε, να μην ε, θεωρηθεί όμως ότι σορευτικά μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις δυνατότητες. Το πλαίσιο έχει γίνει πιο ιεραρχικό, έχει γίνει πιο δίσκαμπτο, έχει γίνει πιο ανώνυμο σε επίπεδο διαχείρισης. Πολλές φορές οι υπεύθυνοι αλλάζουν συχνά ρόλους, λένε διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι μία υποχρέωση της ΕΑΤΣΕΑ που δεν έχει καθορίσει πλήρως τον τρόπο λειτουργία της ε, πρέπει να δώσει περισσότερες δυνατότητες στους ε, αρμόδιους να γνωρίζουν και το οργανόγραμμα κατά τομέα. Έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή μια ιεραρχική σχέση ε, πάρα πολύ δίσκαμπτη. Δεν λειτουργούν οι επικοινωνίες μεταξύ των διαφόρων ταμείων, τα λεγόμενα desk δεν έχουν τις σωστές σχέσεις με τη Γενική Διεύθυνση και με το σύνολο της υπηρεσίας. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα με το Μέντια και λιγότερο καλά με το θέμα του προγράμματος Κουλτούρα. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει και με τους εταίρους της στρατηγικής ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στην εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι θα έλεγα τα αιτήματα αυτών που δεν έχουν επιλεγεί. Θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο όπως έλεγα πριν τα δέσκα να γνωρίζουν καλύτερα το θερμόμετρο της κατάστασης των προγραμμάτων και των αιτημάτων στις διάφορες χώρες. Ε, έχουν ένα σύστημα το οποίο ονομάζουν NING και νομίζω ότι δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στο ε, τέτοιου είδους υποβολές προγραμμάτων ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η χρηματοδότηση όταν επιλεγούν δεν είναι πολύ ικανοποιητικός. Υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία ή εκθέσεις ή τακτικές ε, δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, δεν αναγνωρίζονται στοιχεία δαπανών. Δεν λειτουργεί το σύστημα όπως λειτουργεί κάπως καλύτερα σε προγράμματα όπως το Horizon 2020. Ε, δεν μπορούν να δημιουργηθούν έτσι σχέσεις και ανάμεσα σε διαφορετικούς Τώρα οι αξιολογήσεις των εμπειρογνωμόνων γίνεται θα έλεγα από απόσταση. Γνωρίζω βέβαια τα όρια τα οποία υπάρχουν και τους περιορισμούς στον τομέα της μετακίνησης κτλ. Αλλά τώρα ένας σε μία χώρα, ένας άλλος σε άλλη χώρα, δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλο και αξιολογούν με διαφορετικό φυσικά τρόπο ένα συγκεκριμένο έργο, μια συγκεκριμένη πρόταση, δεν συναντώνται ποτέ και αυτό δημιουργεί προβλήματα και αποκλίσεις. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς ε, υπάρχει και στο Horizon, χειροτερεύει η κατάσταση και στο Horizon. Είναι σαφές ε, ότι το Skype εδώ δεν αρκεί. Προτιμώνται λοιπόν κάποια προγράμματα τα οποία είναι απλά καινοτόμα και δεν εμβαθύνουν οι εμπειρογνώμονες στην πραγματικότητα της κάθε χώρας. Πιστεύω λοιπόν ότι το Creative Europe είναι ένα πάρα πολύ απαραίτητο πρόγραμμα. Έχει αρκετές δυνατότητες αυτοβελτίωσης, έχει προβλήματα διαχείρισης και αναφέρομαι στο ΑΣΕΑ, ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ειδωθεί σύντομα. Πιστεύω επίσης ότι είναι απαραίτητο να πετύχουμε τον στόχο της καλύτερης κυκλοφορίας των δημιουργών, των έργων τους σε επίπεδο οπτικο-ακουστικό, να διεθνοποιήσουμε τις σταδιοδρομίες και να λειτουργήσει το σύστημα αυτό ε, πιο ανταγωνιστικά έτσι ώστε να μπορεί να εξάγεται αν θέλετε και καλύτερα. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας, προβλήματα γραφειοκρατικά, προβλήματα διαφάνειας, προβλήματα χαμηλής εμπλοκής των ιδίων των εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού. Ε, στην επταετία λοιπόν 21-27 θα έχει διευρυνθεί, αν θέλετε, το χαρτοφυλάκιο αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει μια ξεχωριστή γραμματεία για την κουλτούρα, να υπάρχουν επίσης πιο εγκάρσιες μορφές συνεργασίας. Ε, το Horizon ασχολείται περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν με την πολιτιστική κληρονομιά, παρά με θέματα όπως η ε, πολιτιστική διπλωματία. Νομίζω όμως ότι διατηρώντας καλύτερα την κουλτούρα σαν βασικό υποπρόγραμμα, και αυτό είναι μια δική μου αντίληψη αν θέλετε που σας προτείνω, θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες αυτόνομες δράσεις στο πλαίσιο των υποπρογραμμάτων και για τις ε, δημιουργικές οικονομικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικές κτλ και το άλλο αφορά τις ε, τρίτες χώρες. Αυτά είναι θέματα ε, στα οποία θα πρέπει να γίνει κάποιος διάλογος από εδώ και πέρα σε σχέση με το Creative Europe. Υπάρχει θέμα και με τη νομική βάση, το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτό θα δείξει αν μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα προϋπολογισμό ε, χαμηλότερο ή μάλλον υψηλότερο από αυτό το 0,4%. Σε επίπεδο χρονισμού τώρα, μετά από τις καινοτομίες των τομέα των οικονομικό, ε, στις 5 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει η παρουσίαση των μελετών ε, Εκεί θα υπάρξουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, θα υπάρχει δυνατότητα για συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και πέρα από αυτό στις 25 λοιπόν Σεπτεμβρίου θα κατατεθούν οι μελέτες. Έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν. Και η σημερινή συνάντηση θα είναι μια πρώτη συνάντηση επαφής. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι το στοιχείο καινοτομία πάνω στο οποίο θα έλεγα πρέπει να σταθούμε λίγο. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε στο παρελθόν. <clears throat> Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σιμάνοβιτς. και μετά θα πάρουν το λόγο οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση του που βρισκόμαστε τώρα και, τι, και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την ε, εφαρμογή της διευκόλυνσης εγγύησης ε, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα εργαλείο του Creative Europe, για τους στόχους του Creative Europe, για την χρηματοδότηση των κλάδων αυτών, γιατί ε, επλήχθησαν από τι περικοπές. Άρα υπέγραψε την τελευταία μέρα του Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σχετική συμφωνία και ξεκίνησε μια δραστηριότητα για την επικοινωνία. Ανακοινωθέντα τύπου ερωτήσεις ε, συχνές που περιγράφουν το πρόγραμμα αυτό και έτσι το Creative Europe Desk μπόρεσε να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα αυτά αναχώρα. Το ίδιο ισχύει και για τι τράπεζε με τις οποίες ε, ε, επικοινώνησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Γιατί το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή του προγράμματος που ξεκινάει με τη δημοσίευση των ε, αιτήσεων ε, για την υποβολή προσφορών. Και αυτά λοιπόν θα δημοσιευθούν όλα τις επόμενες ημέρα, Υπέρες. Αυτό που είναι σημαντικό στο σημείο αυτό είναι ότι όταν δημοσιευτούν αυτά τον Ιούλιο του 2016 θα ξεκινήσει η διαδικασία, θα είναι ανοιχτή η διαδικασία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Άρα υπάρχει πολλή χρόνο για τους οικονομικούς διαμεσολαβητές στις διάφορες χώρες να αναλυθεί το κατά πόσον το πρόγραμμα του ενδιαφέρει και αν θέλουν να υποβάλουν αίτηση. Μετά τη δημοσίευση λοιπόν που ακολουθεί την νομική βάση του Creative Europe θα στέλνουν οι τράπεζες τις αιτήσει τους για τους πολιτισμικούς κλάδους και τα δημιουργικού κλάδους που θα καλύψει κάποιες από τις βασικές ανάγκες των επιχειρήσεων όπως είναι οι επενδύσεις, κάποια δάνεια γέφυρες και το καθεξής. Οι αιτήσει αυτές θα περάσουν από έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τη σχετική αντιπροσωπεία και θα υπογραφεί η Συμφωνία Εγγύησης που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει η υλοποίηση του εργαλείου. Και από την στιγμή αυτή, φαντάζομαι ότι αυτό σε κάποιες χώρες θα μπορούν να γίνει και από το 2016 ήδη, θα ξεκινήσουν τα δάνεια για τις οργανώσεις και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον πολιτισμικό κλάδο και τον κλάδο τον δημιουργικό. Το δεύτερο εργαλείο είναι το capacity building η τεχνική αρρωγή για τους οικονομικούς διαμεσολαβητές. Αυτό ως σκοπό έχει να διαλευκάνει τις ανάγκες των επιχειρήσεων από τον κλάδο αυτό. Με τόσο συγκεκριμένα λοιπόν εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και σωστή επικοινωνία. Όχι μόνο για να εξηγήσουμε στα εργαλεία τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα εργαλεία αυτά, αλλά για να κάνουμε και τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν την ευκαιρία αυτή να βελτιώσουν τις δραστηριότητες τους, να τις αναβαθμίσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ταμείο Επενδύσεων, ενημερώνει τις διάφορες ιστοσελίδες. Υπάρχει πληροφορία στο, πληροφορία στην ιστοσελίδα του Creative Europe. Και θα τονίζεται και η πρόσβαση τη χρηματοδότηση στις ιστοσελίδες αυτές. Αυτό γίνεται και σε όλες τις ιστοσελίδες για τα οικονομικά μέσα και επίσης θα, τρο, θα προβληθεί και στο, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Έχει γίνει ήδη και μια δραστηριότητα ενημέρωση του κοινού. ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιο συνήθει ερωτήσει για του δικαιούχου και σκοπεύουμε όλα αυτά να τα δημοσιεύσουμε μετά τι θερινέ διακοπέ. Αυτό είναι ο σκοπό μας. Ένα εγχειρίδιο επίση, ένα φυλάδιο, το οποίο θα διατίθεται σε όλες τις ε, γλώσσες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να το μοιράσει λοιπόν σε όλε τι χώρες το Creative Europe Desk. Επίση, ε, υπάρχει και ένα πίνακα για τους οικονομικούς δημοσιολαβητέ. Τώρα, μας, είμαστε σε συχνή επαφή με τα Creative Europe Days για την διοργάνωση εθνικών ημερίδων ενημέρωσης και τέτοιες ε, αιτήσει έχουν έρθει και από τη Γερμανία και από τη Ρουμανία προς το παρόν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα το πώς λειτουργούν όλα αυτά. Να αναφέρω το Ευρωπαϊκό ε, Γραφείο στην ε, Βενετία, με την Biennale της Βενετίας. Ξέρετε ότι έχει πολύ ε, μεγάλο αντίκτυπο η Biennale ως εκδήλωση. Και αυτό θα μπορούσε να ενδιαφέρει και τις τράπεζες της περιοχής, αλλά και οργανώσεις που καλύπτουν μια σειρά δραστηριοτήτων, γιατί το εργαλείο αυτό ουσιαστικά έχει νόημα μόνο αν καλύπτει ε, διάφορους τομείς πολιτισμικούς. Επίσης, το Μποζάρ προετοιμάζεται μια δραστηριότητα για να καταγραφεί το πώς τα νέα οικονομικά μέσα τα οποία είναι εντελώς καινούργια στην αγορά και κατά πάσα πιθανότητα είναι τα πρώτα ε, είναι τα πρώτα και τα μοναδικά που έχουν τόσο ευρύ αντίκτυπο ε, στον πολιτισμικό κλάδο. Αυτό λοιπόν συζητήθηκε και με τους ε, ενδιαφερόμενους φορεί. Να πω επίσης ότι οι τράπεζες που έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Τομέα Επενδύσεων θα πρέπει να αφιερώσουν μια δική εκστρατεία για τι επιχειρήσεις αυτές στη χώρα τους, στις εταιρείε δηλαδή. Αυτά λοιπόν θα είναι τα ενδεχόμενα αποτελέσματα, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτή είναι η δομή του προπολογισμού. Καταρχάς το 2016 και μόνο θα πρέπει να δούμε και το επίπεδο των προσδοσκιών με 120 εκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι ο όγκος των επενδύσεων θα είναι πάνω από 600 εκατομμύρια. Αλλά χρειάζεται η δέσμευση αυτή, γιατί πρόκειται για δεσμεύσει πληρωμών, όχι πληρωμέ, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μπορεί να υπογράψει τέτοιε συμφωνίε με τράπεζε για να ξεκινήσουν τη δουλειά του. Άρα, έχουμε ξεκινήσει με μάλλον χαμηλά ποσά και θα πρέπει να δούμε και τα επίπεδα των προσδοκίων, να δούμε πόσες ε, τράπεζες θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Και βλέπετε λοιπόν ε, ποια είναι τα μελλοντικά μας σχέδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να διανύμετε σε όλους τους συναδέλφους, κυρίως τους και αλλά όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Πολιτισμού, αυτές τις ε, πληροφορίες ε, ενδελεχώς. Να δούμε αν θα ξεκινήσει η πρόσκληση υποβολή προσφορών στις 16 Ιουλίου, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν τα εθνικά γραφεία συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία ευθύ εξ αρχής. Δηλαδή, αυτά τα γραφεία θα κάνουν αυτές τις εθνικές μέρες ενημέρωσης κατόπιν ετήματος. Εντάξει, το κατάλαβα, αλλά συναντηθήκατε στι Βρυξέλλες με τα εθνικά γραφεία εξηγώντα τη στρατηγική, τι πρέπει να κάνουν. Ε, να ενημερώνονται, διότι τελικώ ενημερώνονται τελευταίοι. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν βελτιώνεται καθόλου η διαχείριση. Δεν αναφέρομαι σε εσά, δεν είναι δική σα ευθύνη. <laughs> Από αυτό που κατάλαβα. Μπορεί να κατάλαβα και λάθος. Όπως εμείς ε, ειλικρινά το, το μαθαίνουμε τελευταίοι, ε, γιατί ανακοινώθηκε και την τελευταία μέρα το μάθαμε. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει λίγο καλύτερη επικοινωνία. Εάν τα εθνικά γραφεία, τα οποία θα είναι τα πρώτα τα οποία θα κληθούν να οργανώσουν πράγματα, ε, οι ενδιαφερόμενοι, οι τράπεζες, τα γραφεία, τα ενημερώσατε εκ των προτέρων όλα αυτά και επίσης πώς τους έχετε εμπλέξει ώστε να έχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε την ημέρα την οποία θα ξεκινήσει η πρόσκληση υποβολίου προφερών να το ξέρουν και να μπορούν να απαντήσουν σε όσους ενδιαφέρονται. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ενός προγράμματος, ε, το οποίο βλέπουμε πόσο πολύ ε, απογοητεύει όσον αφορά τα κονδύλια και πόσα περισσότερα περιμέναμε. Πολύ ωραία η Βενετία, πολύ ωραία να βρεθούμε όλα τα λέμε, αλλά εγώ αναφέρομαι σε κάτι άλλο. Σα ευστώ την προσοχή, πρέπει να είναι σαφής η διαχείριση. Ο μειοδιωτικό διαγωνισμό δεν αφορά μόνο τα οπτικοακουστικά μέσα και δεν αφορά μόνο τι επιχειρήσει. Πρέπει να είναι σαφές σε όλου. Πρώτε και κυριότερες οι τράπεζε, σύστημα δημιουργία ικανοτήτων, ενδιαφερόμενοι. επομένω, η προσφορά ε, καθορίζει τη ζήτηση. Εάν δεν εκπαιδεύεται η ζήτηση να γνωρίζει τι θα μπορέσει να βρει, θα υποβάλουν προσφορέ μόνο για το οπτικοακουστικό. Αν ε, μόνο τη Βενετία, πολύ ωραία. Αλλά ε, θα πρέπει να υπάρχουν και ενδιαφέρον από άλλου ε, και από ε, ε, πολιτισμικές οργανώσεις, μουσεία παραδείγματο χάρη. Καταλαβαίνω ότι η Γενική Διεύθυνση Connect που ήταν αρμόδια να το διαχειριστεί όλο αυτό πρέπει να κάνει κάτι, αλλά δεν μπορεί να είναι απλώ ένα θέαμα όλη αυτή η ιστορία να στρεβλώνουμε απλώς ε, ε, και να ε, μην ενημερώνουμε τους συνομιλητές μας. Τα εθνικά γραφεία πρέπει να συμμετέχουν και τη στρατηγική αυτή πρέπει να την κάνουν κτήμα τους αμέσως. Πρέπει να κάνετε μια συνάντηση με τα γραφεία στις Βρυξέλλες, όχι όταν τους ρωτήσουν θα πάνε. Επίσης δεν φτάνει όλη αυτή η χαρτούρα, αυτή η έκθεση έτσι ψυχρή και ανώνυμη. Χρειάζεται συμμετοχή των εταίρων της Δημιουργικής Ευρώπης και πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ότι οι τράπεζες θα από τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσουν ισορροπημένα χαρτοφυλάκια για ένα πολύ διαφοροποιημένο κόσμο. Για από το μικρό στο μεγαλύτερο, από τι μη κερδοσκοπικέ στι κερδοσκοπικέ. Το ζητήσαμε, εγώ το υπερασπίστηκα ω εισηγήτρια γιατί ήταν έτοιμοι να το κλείσουν το θέμα αυτό. Όταν ξεκίνησε ο κανονισμό. Λοιπόν, δεν θα ήθελα στην πράξη ε, να. Ε, χαθεί ένα εργαλείο που το περιμένουμε τόσο καιρό. Το περιμένουμε δυόμιση χρόνια και τελικά το μαθαίνουμε την τελευταία μέρα και κανένα δεν ξέρει τίποτα. Αυτό αποτελεί παράδειγμα αυτό που σας λέω ότι δεν υπάρχει αίσθηση συνδιαχείριση. Ε, μετά θα μου πείτε ότι τα ξέραν όλα, είναι πλήρως ενημερωμένοι και τα ξέρουν όλα και ότι ξεκινούν τα πράγματα με όλους ενημερωμένους. Εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση. Ε, ε, τα λέω και λίγο παθιασμένα, αλλά νομίζω ότι πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν επί τόπου. Τώρα, πρώτα στο λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Μπέντα, ο κύριος Τζαμπάσκι και ο κύριος Μίκελς και ο κύριος Μόργαν. Όχι, δεν θέλει ο κύριος Μόργαν. Η κυρία Μίκελς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ήδη υποδείξατε ότι είστε ιδιαίτερα δεσμευμένοι και μας δώσατε πολλές πληροφορίες ε, για το πρόγραμμα Creative Europe, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και το καθεξής. Δεν πρόκειται να επισελθώ σε λεπτομέρειες και συζητήσαμε επίσης το θέμα των οικονομικών μέσων. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό θεωρώ είναι τα εθνικά γραφεία σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Creative Europe έχουν θετικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί βοηθούν στην εφαρμογή των όλων αυτών των στοιχείων. Έχουμε και κάποια στοιχεία στη διάθεσή μας, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι χώρες που συμμετέχουν δεν είναι εξίσου αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητε και τις ικανότητες των εθνικών γραφείων που θα πρέπει να ασκούν και ρόλο συντονιστικό για τους ε, αλλά παράλληλα θα πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση και να εντοπίζουν αδεχόμενες ανάγκες των δικαιούχων ε, εγγυήσεις ε, και αντιεγγυήσεις. 21 δισεκατομμύρια για τον προϋπολογισμό, αναφέρθηκε το ποσό αυτό. Όταν μιλάμε για εγγυήσεις πιστώσεων θα πρέπει να αναφέρουμε και το θέμα της ανάπτυξης δυναμικού και οικονομικής οικονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κλάδου του πολιτισμικού. Και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ε, του κλάδου αυτού θα πρέπει να λεφθούν υπόψη. Και δεν μιλάω μόνο για το σύνολο του κλάδου, αλλά και για τις υποενότητες της αγοράς αυτής. Τα οικονομικά λοιπόν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να δίνουν και πληροφορίες σχετικά με αυτό. Οι οντότητε, λοιπόν, οι εταιρείε, οι φορεί που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων όπως το COSME, όπως το ορίζοντα 2020 και συνοψίζοντα θα ήθελα να πω ότι προσβλέπω και στη συνεργασία με την Πρόεδρο και τους συζητητές. ευχαριστώ Η κυρία Μίκελς. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την Πρόεδρο για την ε, μεγάλη και δεσμευσή της. Ε, και σε ό,τι αφορά την ε, ενημερωτική πολιτική και για α, όλους αυτούς που πρέπει να διαβιβάσουν το μήνυμα. Αυτό έχω πέσει σημαντικό ρόλο, ξέρετε, και νομίζω ότι αυτό συχνά αποτελεί ένα σημείο που χωλένουν τα προγράμματα. Και γι' αυτό τελικά σε πολλές περιπτώσεις τα προγράμματα δεν ε, υλοποιούνται με επιτυχία. Δεν θα μακρηγορήσω. Είπατε ότι θα κάνουμε και άλλη ε, ε, εκτενή συζήτηση Χθε είχαμε και την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Βιομηχανία και συζητήσαμε το νέο Ταμείο Εγγυήσεων και θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω ότι η δημιουργική βιομηχανία, ο δημιουργικό κλάδο δεν περιλαμβάνει τα πάντα. Το Creative Europe είναι πολύ πιο ευρύ. Και θεωρώ ότι σε όλα τα οικονομικά μέσα, είτε πρόκειται για πιστώσει, είτε πρόκειται για έμεσε επιδοτήσεις, πάντα τέτοια πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. οι μικρές επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις. Αυτό είναι το θέμα. Και στην ε, βιομηχανία αυτή και στον κλάδο αυτό. Και έτσι το ΕΦΣΥ, το οποίο προβάλλεται ως το κατεξοχήν επιτυχημένο πρόγραμμα, τελικά δεν προωθεί τέτοια δημιουργικά project. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κατανομή των τομέων και των κλάδων, αλλά και η περιφερειακή διάσταση, μάλλον η διάσταση της περιφερειακής ε, διανομής του ΕΦΣΥ. Είναι ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί. Για παράδειγμα, στη δική μου χώρα δεν έχουμε ούτε ένα project από την Ανατολική Γερμανία για το ΕΦΣΙ. αυτό, όπως και να το κάνουμε, μας προβληματίζει. Το Ταμείο, λοιπόν, ύψους 121 εκατομμυρίων. Ε, θεωρώ ότι και σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να δώσει κάποια ε, ενάυσματα, να αλλάξει κάτι. Και ελπίζω ότι και καινοτομικές, ε, δημιουργικές εταιρείες θα υποστηριχθούν και όχι μόνο οι μεγάλες ε, εταιρείε. Έχω αμφιβολίες όμως γι' αυτό. Και όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπορούμε να τα εντάξουμε και στο πλαίσιο των συζητήσεών μας μετά το καλοκαίρι. Και φυσικά θα συμμετέχουμε με μεγάλη χαρά. Ναι, βεβαίως. Ε, θα εμβαθύνουμε και με τους ε, υπευθύνου των ε, μελετών που θα μας κάνουν την παρουσίαση και καλά κάναμε και το να βάλαμε αυτό για τις 5 Σεπτεμβρίου ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Η κυρία Σβεντρόβα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, απαιτείται χρόνος και για τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να υπογραμμίσω όμως κάτι το οποίο αναφέρθηκε από συναδέλφους χτες. Η προετοιμασία των πιστώσεων για το Ευρωπαϊκό Έτος ε, Πολιτισμού. Ε, πιστεύετε ότι θα ετοιμαστούν τα πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουμε με τη σειρά μας να κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Ε, sappiamo che questo... Γνωρίζουμε αγαπητή Σοίντροβα ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, ε, για το οποίο έχουμε δώσει μάχη. Δεν είναι κάτι που έχει σχέση με το Creative Europe και ιδιαίτερα με τον προϋπολογισμό του Creative Europe. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό στην Επιτροπή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να περικόπτουμε κάποιους ασθενείς έτσι και αλλιώς οικονομικούς πόρους πρέπει να βρούμε χρήματα εκτός του Creative Europe ε, που εδώ και ένα χρόνο καλύπτεται από συμπληρωματικές δαπάνες. Πάντως υπάρχουν, ε, συμφωνώ, σχέσεις ανάμεσα στα δύο. Απαιτείται λοιπόν να μπορέσουμε να καλύψουμε την πρόκληση αυτή. Δεν ξέρω αν ο Μόργανο θέλει το λόγο, αφού επιμένεις. Νομίζω ότι το παιχνίδι που παίζεται στην παρούσα φάση είναι αυτό το οποίο συνδέεται με ένα πρόγραμμα το οποίο ως έχει από μόνο του αν θέλετε και αν δούμε πραγματικά τους αριθμούς που έχουμε στην διάθεσή μας σε σχέση με την απασχόληση, σε σχέση με τις μικροεπιχειρήσεις κάτω των εννέα εργαζομένων μας δείχνουν ότι υπάρχει χώρος, σημαντικός χώρος, στον οποίο μπορούμε να κινηθούμε και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να δώσουμε απάντηση στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα του Juncker εδώ, στο πρόγραμμα το οποίο έχει σαν στόχο την οικονομική ανάκαμψη και την απασχόληση των νέων. Τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας μας δείχνουν ότι αυτοί που ασχολούνται με τους συγκεκριμένους τομείς εδώ και πολλά χρόνια θίγονται και δεν υπάρχει κανένας άλλος παραγωγικός τομέας όμως ο οποίος να είναι σε θέση να απορροφήσει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό αυτού του επίπεδου. Η απάντησή μας λοιπόν είναι διπλή και απασχόληση και κυρίως μια απασχόληση υψηλής ποιότητας. Όλες αυτές οι συζητήσεις βέβαια ε, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για να γίνουν πράξη και η πράξη διευκολύνεται από την πρόσβαση στις πιστώσεις και μέσω εγγυήσεων αυτών των ε, ταμείων μέσω των προκαταβολών ίσως και ένα άλλο θέμα είναι ακριβώς ε, ε, η προστασία του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας ακριβώς και της προστασίας ε, των νέων επιχειρήσεων. Εδώ απαιτείται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης και συνδυασμού δυνάμεων, γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι εμένουμε σε κάποιες επιλογές οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια έλλειψη αντικειμενικότητας και που οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν βρίσκονται στο ύψος των δυνατοτήτων που έχει ο τομέας αυτός. Είναι μια πρόσκληση λοιπόν αυτό το οποίο κάνω, άλλωστε και η παρέμβαση της Προέδρου στην αρχή της συνεδρίασης δείχνει νομίζω ε, τις θέσεις τις οποίες όλοι συμμεριζόμεθα για μια επιθυμία του Κοινοβουλίου να ακολουθήσουμε την συγκεκριμένη αυτή πολιτική. Σας ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπαμε πολλά πράγματα, είπαμε πολλά στοιχεία, δώσαμε πολλά στοιχεία. Βρισκόμαστε στην πρώτη, αν θέλετε, συζήτηση. Στις πέντε θα συζητήσουμε και στις 8 Νοεμβρίου θα κατατεθεί η ε, πρόταση της έκθεσης, αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά πριν φτάσουμε σε αυτή τη φάση, για να γνωρίζουμε ποια είναι τα στοιχεία που θέλετε να εμπεριέχονται. Λοιπόν, η Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλημέρα. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την ε, εις βάθος ματιά στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, διότι έρχεται να προστεθεί πολύ καλά στην λεγόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος. Ε, θα υπάρξει μια ενδιάμεση αναθεώρηση και από αυτή την άποψη είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ότι μπορούμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση και ε, μπορούμε να δούμε και τι γίνεται με την εφαρμογή του προγράμματος γιατί αυτό που είναι το πιο σημαντικό για μας είναι να έχουμε ότι καλύτερο μπορούμε από αυτό το πρόγραμμα και να έχουμε ένα πρόβλημα υψηλής ποιότητας στο δεύτερο τμήμα της εφαρμογής. Είμαστε πλέον 2,5 χρόνια μετά από την έναρξη του προγράμματος που σημαίνει ότι έχουμε περάσει διάφορες αναταραχές και αλλαγέ. Αναφέρθηκε ότι το πρόγραμμα ε, χωρίστηκε διοικητικά μεταξύ δύο γενικών διευθύνσεων και δύο επιτρόπων και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε μαζί με τους αδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Connect ότι το, πρόβλημα, το πρόγραμμα θα παραμείνει ακέραιο, ότι θα ε, τηρήσουμε τα όσα αναφέρονται στη νομική βάση του προγράμματος. Ε, υπάρχει μια task force, μια ομάδα ειδικών καθηκόντων που καθορίζει τα διάφορα στοιχεία. Ε, διαχειριζόμαστε μαζί τα διακλαδικά στοιχεία, ενημερώνουμε αλλήλους για το τι ακριβώς γίνεται από την πλευρά του media και τι γίνεται από την πλευρά του culture και φυσικά προσπαθούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα. Νομίζω ότι προς το παρόν η διαχείριση του προγράμματος ε, διασφαλίζεται από τις δύο γενικές διευθύνσεις και από τους δύο επιτρόπους παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα διοικητικό κενό. Τώρα, όσον αφορά την πολιτιστική πλευρά του προγράμματος, καθήκον μας είναι να διατηρήσουμε την πολιτισμική πολυμορφία στην Ευρώπη, να υπάρχει ανταγωνιστικότητα των πολιτιστικών επιχειρήσεων και να υπάρχει κινητικότητα των όσων συμμετέχουν σε πολιτισμικά δρόμενα στην Ευρώπη και φυσικά ε, κατ' εξίσου σημαντικό να προωθήσουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο ο οποίος φυσικά είναι πολύ πιο σημαντικός αυτή τη στιγμή από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ε, δεδομένων και των τελευταίων εξελίξεων με τους πρόσφυγες ε, στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα ανάλογα με τις ε, ε, ανάγκες που ανακύπτουν και τις δυνατότητες που μας προσφέρει φυσικά η, η νομική βάση. Βάσει των δυνατοτήτων αυτών μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα λογικό μείγμα ε, ώστε να υπάρχει συνέχεια, δηλαδή αυτά που κάναμε στο πρόγραμμα κάλυψης στο παρελθόν και καινοτομίας, δηλαδή νέα στοιχεία, νέες προσεγγίσεις, ε, να μπορούμε να σκεφτόμαστε χωρίς στεγανά και να υπάρχουν πραγματικά καινοτόμα προγράμματα. Όσον αφορά το πολιτισμικό σκέλος του προγράμματος, πιστεύω ότι ε, τα καταφέρνουμε μόνο μέσω προγραμμάτων συνεργασίας. Ε, η σύνθεση αυτών των προγραμμάτων από Τη δική μας τη σκοπιά αντανακλά αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, παρά το γεγονός ότι ε, μπορεί να υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση ε, των... το θέατρο, το κινηματογράφο κλπ. σε σχέση ε, με τα υπόλοιπα είδη. στο τμήμα του προγράμματος που αφορά ε, το ε, Media θα έχουμε την τελευταία πρόσκληση υποβολής προσφορών ε, στο τέλος του έτους και στα επόμενα τέσσερα χρόνια που θα διαρκέσει το πρόγραμμα θα μπορέσουμε, ελπίζουμε να έχουμε ένα κατάλογο δικτύων τα οποία θα εκπροσωπούν όλα στους σημαντικούς πολιτισμικούς τομείς και υποτομείς στην Ευρώπη και και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα θα αποτελούν αξιόπιστο εταίρο, διότι θα είναι μια εικόνα της κατάστασης σε όλη την Ευρώπη για θέματα πολιτισμού. Στο υποπρόγραμμα λοιπόν Culture ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μεγάλες οργανώσεις στην Ευρώπη οι οποίες βασίζονται σε ανερχόμενους ε, καλλιτέχνες, να υποστηρίζουν τους νέους καλλιτέχνους παντού στην Ευρώπη και να μπορέσουμε να έχουμε ευρωπαϊκό προγραμματισμό σε όλα. Υπάρχει πολύ καλή εμπειρία με τις 8 πλατφόρμες που έχουμε συστήσει μέχρι τούδε και ελπίζουμε ότι στις αρχές του επομένου έτους θα μπορέσουμε να πούμε ότι τους έχουμε διπλασιάσει και θα συνεχίσουμε με αυτό το σκοπό και κυρίως ε, θα ανταποκριθούμε και στη δική σας την επιθυμία ε, έχουμε τρεις ε, προσκλήσεις υποβολή ε, προσφορών σε μία επταετία. Αυτή θα είναι η τελευταία πρόσκληση και ελπίζουμε ότι θα διασκεδάσουμε και τη δική, <laughs> τη δική σας την ανησυχία. Δεν θα είναι μόνο οικονομική προσέγγιση, αλλά θα έχουμε και καλλιτεχνικές και ε, άλλες αντιστοιχίες όσον αφορά το δίκτυο των γραφείων Creative Europe που αναφέρθηκε. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τα εθνικά γραφεία και μάλιστα για ένα τόσο μικρό πρόγραμμα είμαστε και ευτυχείς που υπάρχει αυτό το δίκτυο. Δεν ήταν εύκολα βέβαια τα πράγματα σε κάποιες χώρες να συγχωνευτούν τα γραφεία, το πρώην ε, ε, σημείο επαφή για το culture και το σημείο επαφή για το media που τώρα έχουν γίνει ένα δίκτυο. Αλλά μετά από δύο χρόνια πρέπει να πω ότι στο 99% των περιπτώσεων λειτουργεί σχεδόν καλά το ε, σύστημα και οι συνάδελφοι που εργάζονται στα εθνικά γραφεία ε, χαίρονται για τη συνεργασία. Έχει βελτιώσει την κατάσταση και για αυτούς, διότι έχουν γίνει πιο ισχυροί μέσω αυτής της συγχώνευσης και για μας φυσικά αυτό είναι ένα πάρα πολύ ε, πολύτιμο δίκτυο. Του συναντούμε δύο φορές το χρόνο και φυσικά υπάρχουν και ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα μόνιμης επικοινωνίας με τα γραφεία αυτά και πρέπει να δούμε και την έκθεση που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε τι ελλείψεις υπάρχουν, ε, διότι αναφέρατε κάποιες ελλείψεις. Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα, έγιναν δύο ε, σεμινάρια εκπαιδευτικά για τα γραφεία, για τα χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάμε περαιτέρω. Ε, τα γραφεία είναι πλήρως εξοπλισμένα, αλλά δεν ξέρουμε πού θα ξεκινήσει το μέσο πρώτα, σε ποια χώρα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε φρούδες ελπίδες και να είναι διαθέσιμο το μέσο σε δύο χρόνια και εμείς να τους πούμε ότι θα είναι τώρα. Όταν θα ξέρουμε από πού θα ξεκινήσουμε, φυσικά θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί και θα ε, φροντίσουμε να το διαβιβάσουμε και να υπάρχει και σχετική επικοινωνία. Κάτι τελευταίο για τις τρίτες χώρες. Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε χώρες της ε, ανατολικής και νότιας γειτονίας. Συνεργαζόμαστε με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία ήδη. Και υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον. Έχουμε ξεκινήσει διαπραγμάτευση και με την, την και το Ισραήλ. Έχουν προχωρήσει αρκετά οι διαπραγματεύσεις, αλλά φυσικά υπάρχει το μεγάλο πρόσκομα της νομικής βάσης διότι πρέπει να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση της νομοθεσίας με την οδηγία EVMS, που είναι η προϋπόθεση συμμετοχής στο υποπρόγραμμα Media. Πρόκειται για μία από τις επιπλοκές φυσικά για αυτές τις χώρες ε, και δεν μπορούν να συμμετέχουν ε, στο πρόγραμμα, αλλά μπορούν σίγουρα να συμμετέχουν στο τμήμα του Culture παρατηρήσεις που ακούστηκαν ε, για τη διοικητική διαχείριση του προγράμματος, αιτήσει και το καθεξής. Αυτά θα τα αφήσω να σας τα πει ο Μπράιαν, που είναι και ο αρμόδιος. Και ξέρει τα, της καθημερινής διαχείρισης του προγράμματος. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα στείλουμε τον Οκτώβριο μια αντιπροσωπεία στην Τινησία και καλό θα είναι μέχρι τότε να έχουμε κάτι να μεταφέρουμε. Οι σχέσεις με το Μαρόκο, την Τινησία είναι εξαιρετικέ. Έχουμε πολλές ε, μονάδες ευρωπαϊκές σε συνεργασία μαζί τους. Ε, συμμετέχουν σε φεστιβάλ κινηματογράφου, πολιτισμού κτλ. Έχετε το λόγο. Όπω και η Κάρλ και εγώ σα ευχαριστώ που μα καλέσατε εδώ σήμερα για τη σημαντική αυτή συζήτηση. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε ο Κάρλ. Νομίζω ότι συμφωνώ και με όλα όσα είπε. Να κάνω όμω κάποια συμπληρωματικά σχόλια θα ήθελα. Σε ό,τι αφορά τη συνδιαχείριση των προγραμμάτων από την DGR και την DG Connect, νομίζω ότι ένα από τα πλεονεκτήματα μεταξύ άλλων είναι ότι βοηθάν τα προγράμματα να έχουν επίδραση και να διαδοθούν και σε άλλους κλάδους σχετικούς ε, από το DJR, για παράδειγμα, μπορούμε να πάμε στην Age 2020. Ε, νομίζω λοιπόν ότι στην DG Connect έχουμε τη νέα Γενική Διεύθυνση για τα Μέσα Ενημέρωση 1η Ιουλίου και ο κ. Μπαμούντα είναι ο Γενικός Διευθυντής. Στην, ε, γενική, λοιπόν, στη Διεύθυνση λοιπόν αυτή έχουμε και μια, ένα τμήμα το οποίο είναι αφιερωμένο στην έρευνα για τις τεχνολογίες μέσων. Και προσβλέπουμε στην αξιοποίηση των συνεργειών αυτών. Σε επίπεδο πολιτικής τώρα. Όπως ξέρετε, ασφαλώς μία από τις προτεραιότητες της θετίας αυτής είναι η νέα ψηφιακή αγορά. Και υπάρχει εδώ μία ρυθμιστική διάσταση σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του copyright, αναθεώρηση των υπηρεσιών των απτοκοστικών μέσων και πιστεύουμε ότι ο κανονισμός δεν φτάνει για να αλλάξει η πραγματικότητα θα πρέπει να υπάρχουν και εργαλεία μέσα τα οποία θα δίνουν ενάψματα και κινήτρα θα βοηθήσουν τον κλάδο να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις ε. και έχουμε και ένα πρόγραμμα για τα μέσα μέσα στο Creative Euros και πιστεύουμε ότι αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για να χρηματοδοτηθούν ε, στις επιχειρήσεις τέτοια μέτρα της μεταρρύθμισης. Ξέρουμε πώς είναι ο οπτικοστικός ε, κλάδος στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αλλάζει. Όταν ξεκίνησε το Creative που που δεν υπήρχε το Netflix καν στην Ευρώπη. Και πλέον αυτό αποτελεί την πραγματικότητα σε όλες μας τις χώρες. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόσφορα και πολύ κοινοτομική και αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση για τους παρόχους της Ευρώπης. Ένα παράδειγμα για το πώς αλλάζουν τα πράγματα και πόσο γρήγορα αλλάζουν κυρίως. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτή η συμπληρωματικότητα με την ψηφιακή ενιαία αγορά αποτελεί ένα βασικό θέμα του προγράμματος, ε, υποπρογράμματος για τα μέσα. Σε ό,τι αφορά τα γραφεία, σύμφωνο και πάλι με τον Κάραλο ότι πρόκειται για ένα στρατηγικό ε, πλονέκτημα για την εκστρατεία αυτή για να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε και να επικοινωνήσουμε. Ιδιαίτερα καινοτομικά στοιχεία. Είτε πρόκειται για το Guarantee Facility που αποτελεί τη βασική καινοτομία ή το σύστημα διανομής online που είναι κάτι διαφορετικό από την υποστήριξη προς τις ταινίες, τους κινηματογράφους κτλ. Η κοινότητα των δικαιούχων σε ό,τι αφορά το βίντεο on demand και τους σχετικούς παρόχους είναι τελείως διαφορετική. Γι' αυτό λοιπόν Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα γραφεία για να μας βοηθήσουν να έχουμε επαφή με την ε, ομάδα αυτή των ε, νέων συσταθήσεων επιχειρήσεων. Θα λάβουμε υπόψη επίσης τα σχόλιά σας και τις ε, παρατηρήσεις σας σε σχέση με όσα παρατηρήσατε και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και πρόκειται για διαφορετικού είδους υποστήριξη. Είναι διαφορετικό το είδος. Περνάμε από τις επιδοτήσεις σε ε, συστήματα υποστήριξης της αγοράς και θα πρέπει να δούμε ε, πώς αυτό, πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο γι' αυτό. Κάποια τέτοια στοιχεία όμως δεν υπάρχουν για τον καραντίο. Facility. Κατανοώ ότι έχετε την αίσθηση ότι έχει περάσει πολλής χρόνος και για μας έχουν περάσει δύο χρόνια. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το τι, ποιος είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε δύο χρόνια. Αλλά είμαστε σε μια πρώιμη φάση ακόμα που θα αποφασίσουμε μαζί με το EIF ποιες τράπεζες θα συμμετάσχουν, από ποιες χώρες και αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε πιο συγκεκριμένη επικοινωνία και ενημέρωση των γραφείων. Να αναφέρω το θέμα και των δικτών, το οποίο θίξατε. Πιστεύουμε, και αυτό σχετίζεται και με το θέμα του προπολογισμού, θεωρώ στενά. Γιατί το προπολογισμό σημαίνει και υποβολή εκθέσεων και συγκεκριμένα αποτελέσματα, από ξέρετε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο πολλές ε, εκθέσεις, αναφορές, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που πετυχαίνει το πρόγραμμα και η ενδιάμεση αναθεώρηση θα μας βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης θέλουμε να συμπληρώσουμε τους υφιστάμενους δείκτες ε, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία. Θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και θα κάνουμε κάποιες τέτοιες προτάσεις. Δεν θα αποφασίσω εγώ προφανώς από θεσμική άποψη ποιε θα είναι οι μελλοντικέ τοποθετήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί προφανώ θα υπάρξει και μία ε, φάση δημοσιονομικού, δημοσιονομικής ε, διαβούλευσης και δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων. Και φυσικά είναι μεγάλε οι προκλήσει, πολλές είναι οι αλλαγέ που σημειώνονται και όσο πιο πολύ υποστηρίξουμε τον κλάδο, τόσο το καλύτερο και για νέου είδου μέσα, τα οποία θα πρέπει δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί, θα αναπτυχθούν και θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες κτλ. Αυτά, ευχαριστώ. Ε, ε, Σας ευχαριστώ. Πάνω στο ίδιο σημείο θα έλεγα ότι έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε μιας και έχει προηγηθεί η συνάντηση που είχαμε με την DG Connect Είχαμε κάνει μια πρόταση σε σχέση με το χρηματοδοτικό μέσο να ενσωματωθεί μέσα στο ΕΦΣΥ. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο για το μέσο αυτό, το οποίο είναι σχετικά περιορισμένο, να αποκτήσει μια νέα φιλοδοξία διάσταση αν θέλετε, να ενώσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή του με αυτά του ΕΦΣΥ και να συνοδεύεται αν είναι δυνατόν από κάτι το οποίο επαναλαμβάνω σε ένα βαθμό δεν συνδέεται άμεσα με το Creative Europe αλλά είναι ένα μέσο αν θέλετε με τις επιχειρήσεις οι οποίες πολλές φορές είναι μικροεπιχειρήσεις και οι οποίες δεν γνωρίζουν με ποια πλατφόρμα να συνεργαστούν. Νομίζω ότι ένα ενσωματωμένο στο ΕΦΣΙ πρόγραμμα θα μπορέσει να διαδοθεί καλύτερα και να είναι ε, πιο ενημερωμένες οι μικροεπιχειρήσεις και επιχειρήσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα μπορούσαμε τα δύο πράγματα αυτά να τα κάνουμε μαζί. Θα δούμε ακριβώς ε, τι δυνατότητες υπάρχουν, τι πιστοτικά ιδρύματα συμμετέχουν και θα αποκτήσουμε μια κρίσιμη μάζα εδώ, διότι ε, για το ΕΦΣΙ μέχρι τώρα για πολιτισμό δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Λίγα πράγματα για την εκπαίδευση και πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε προληπτικά. Αυτό νομίζω έχει άμεση σχέση με την στρατηγική που θα ακολουθήσετε και εσείς σαν Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο τώρα λοιπόν τον Διευθυντή της ΑΤΣΕΑ. Χαίρομαι που είναι μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τα στοιχεία και τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ κυρία Κώστα. Χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να παρουσιάσω την εφαρμογή του προγράμματος. Νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου για να βοηθήσουμε τα desk να λειτουργήσουν. Έχουμε δημιουργήσει μια κοινότητα online χρησιμοποιώντας τα αγγλικά όπως είπατε. Θα πρέπει να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες μας καλύτερα στις 26 Οκτωβρίου θα έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση για το πώς θα βελτιώσουμε τις σχέσεις αυτές και πριν τη συνάντηση αυτή να δούμε τι πληροφορίες και ενημέρωση μπορούμε να κάνουμε. Είπατε ότι τα ΔΕΣΚ θα ήθελα να είχαν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις αιτήσει, ιδιαίτερα όταν απορρίπτονται αυτές οι αιτήσει. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι πληροφορίες μπορούμε να παρέχουμε σαν Επιτροπή. Υπάρχει βέβαια το θέμα εδώ της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να ζητάμε αν θέλετε και την έγκριση αυτών που ζητούν να γίνει δεκτό το πρόγραμμά τους να μεταφέρονται τα στοιχεία τους στα desk. Σε σχέση με τον χρονισμό μπορούμε να ενημερώσουμε τα desk. Αυτή τη στιγμή ληφθούν οι αποφάσεις βέβαια. Δεν είναι άμεσο ίσως, ε, δεν είναι δυνατό να ενημερώνονται την ίδια στιγμή, αλλά παρόλα αυτά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε όπως κάνουμε με το Erasmus+ και τις Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης. Στο παρελθόν έπρεπε οι αιτήσει αυτές να γίνονται online, χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά έγγραφα, αλλά έχουμε ελαχιστοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, δεν υπάρχει τώρα τέτοια ανάγκη να υποβάλει κανείς και online στοιχεία και μέσω επιστολών παραδοσιακών. Σχετικά με τη χρήση των εμπειρογνωμόνων τώρα, και η συνεργασία των εμπειρογνωμόνων online από απόσταση. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών που κάναμε, εμένοντας το θέμα της ποιότητας βέβαια. Έχουμε μια μεγάλη εμπειρία μέχρι τώρα από τη χρήση των εμπειρογνωμόνων online Πέρυσι κάναμε μια έρευνα με όλους τους εμπειρογνώμονες, κάποιοι από αυτούς είχαν ενημερωθεί online, κάποιοι από αυτούς είχαν έρθει στα γραφεία μας και το 94% είπαν ότι είχαν τις πληροφορίες για να κάνουν τις σωστές αξιολογήσεις. Υπήρξε μια δυνατότητα για τους εμπειρογνώμονες να μετακινούνται, αλλά αυτό ε, γίνεται για να μπορούν να συναντηθούν, να δημιουργήσουν δικτυώσεις, να ανταλλάξουν προγράμματα για το μέλλον. Πάντως είδαμε εμείς ότι σε σχέση με την ποιότητα της αξιολόγησης αυτό δεν ήταν η βασική ανησυχία. Απλά τους άρεσε να συναντώνται μεταξύ τους και να δικτυώνονται. Ε, εμείς κάνουμε online και τα briefing και τις ατομικές αξιολογήσεις και σε σχέση τώρα με κάποια ευαίσθητα θέματα που είναι στο τσάκ ας πούμε για τη χρηματοδότηση. Εκεί που υπάρχουν διάφαρες έχουμε μια άλλη ομάδα εμπειρογνωμόνων στις Βρυξέλλες. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα ίσως που πρέπει να αποφασίσετε με διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες που μπορείτε να μας δώσετε θα μας ικανοποιήσουν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλε ερωτήσεις. Έχουμε μείνει και τρεις και ο κούκο. Θα ήθελα να εμβαθύνω στο εξή. Εγώ θα ήθελα περισσότερα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά αυτού του μέσου. Καταλάβαμε το χρονοδιάγραμμα, πότε θα ξεκινήσει και τα συναφή, αλλά δεν μου δώσατε ειλικρινά λίγο πιο λεπτομερείς πληροφορίες ε, για την κατάσταση. Ε, κάτι ακόμα, μπορεί να μην κατάλαβα και καλά. Εσείς ξεκινάτε το μειοδοτικό διαγωνισμό, υπάρχει πρόσκληση υποβολής προσφορών για όλη την Ευρώπη, για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες κλπ, όχι μόνο τράπεζες όπως είπαμε, και θα εξαρτηθεί από το τύπο των προτάσεων που θα κάνουν, εάν θα ε, ε συμπεριληφθούν στους υποψηφίους και πώς θα λάβετε υπόψη σε αυτό που έχουμε και στον κανονισμό, να υπάρχει και μια γεωγραφική ισορροπία και τομεακή ισορροπία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το περιλαμβάνει ήδη ρητά ο διαγωνισμός. Ήθελα λίγο πιο τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί αυτά τα οποία μάθαμε σήμερα ε, ήταν ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν μα είπατε πράγματα περιεχομένου. Εγώ τη διάβασα τη συμφωνία και ίσω θα μπορούσατε να μα δώσετε και κάποια στοιχεία επιπλέον. Έχουμε μείνει και ελάχιστοι βέβαια, το αντιλαμβάνομαι, αλλά θα ήθελα για την επόμενη συνεδρία σα στις 5 Σεπτεμβρίου να μα δώσετε πιο αναλυτικέ πληροφορίε. Δεύτερον, Κατάλαβα καλά, έτσι. Υπάρχει ένας γενικός διαγωνισμός, μένει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής προσφορών, ωραία, θα υπάρξει ένα κατάλογος κλπ. Τρίτον, είναι σαφέ ότι πρέπει να είναι ισορροπημένο το χαρτοφυλάκιο, να έχουμε του διάφορου ε, ε τομεί κλπ. Εγώ θα ήθελα και γεωγραφική ισορροπία, να μην κερδίσουν στο τέλο οι τράπεζε μόνο μια χώρα, γιατί τελικά ξεχνάμε τη δυνατότητα για του υπολείπου να μπορούν να συμμετέχουν. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφέ. Αυτή η ανησυχία λοιπόν που έχουμε συμπεριλάβει στον κανονισμό, δεν ξέρω καλά με ποιο τρόπο, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια του περιεχομένου του διαγωνισμού. Αυτό για τον κανονισμό και για οτιδήποτε και όχι για άλλο λόγο, συγγνώμη. Μπορεί να χρειάζεται να υπάρχει και ε, συνδυασμός με τα ταμεία του Ταμείου, ε, του ταμείου Στρατηγικού Ταμείου Επενδύσεων ε, του ΕΦΣΥ για να μπορέσουμε να έχουμε κατάλληλη χρηματοδότηση. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτός είναι συνδυασμός των ε, ευκαιριών για τη συνεισφορά κλπ. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να συνεχιστούν και να έχουμε και περισσότερους πόρους σε σχέση ε, με τα όσα έχουμε, να έχουμε συγχρηματοδότηση. Αυτό πρέπει να είναι σαφές δεν ανοίγουμε μια γραμμή προπολογισμού και ξεχνάμε την άλλη. Η άλλη πρέπει να καλύπτει πράγματα που αφορούν ε, περισσότερο τον πολιτισμό, ε, τη συλλογική διάσταση κλπ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Κάτι τελευταίο προς την ε, Ατσέα. Εσείς μας είπατε ότι όσον αφορά τη στρατηγική συμμετοχή των γραφείων μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Το εκτιμώ ιδιαίτερα ότι είστε ανοιχτό και κάνουμε μια πραγματική συζήτηση εδώ. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί κάνει καλό σε όλους. Το σύστημα θα βγει κερδισμένο διότι θα νιώθουν ότι συμμετέχουν και αυτοί στη στρατηγική. Η ερώτησή μου. Όλοι είπαν ότι αυξήθηκε το άχθος και δεν μειώθηκε πρόσβεση, τεκμηρίωση κλπ. κλπ. Και η απλούστευση έμεινε όνειρο μακρινό. Και εσείς λέτε ότι τα ζητάνε μόνο διαδικτυακά και αυτοί λένε ότι πρέπει να έχουν και τεκμηρίωση σε χαρτί και διαδικτυακή. Ε, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μα λένε και όλοι ψέματα. Αλλά κάτι ακόμα. Για τους περισσότερους αυτό είναι μια γκυλοτίνα. Καταλαβαίνω ότι είναι χρηματοδημοτικό μέσο. Αλλά μπορούμε να βρούμε ένα διαφορετικό σύστημα. piccoli e associativi è un disastro e finisce che non... Να μπορούν να έχουν ε, χρηματοπιστωτική πίστη ε, να τους δίνονται δανειοδότηση γιατί περισσότεροι ε, από τους μικρούς λένε ότι είναι μια καταστροφή η όλη διαδικασία και δεν μπορούν να λάβουν δανειοδότηση. Η Γενική Διεύθυνση Connect, όταν λαμβάνει υπόψη τη και αρχίζει να ασχολείται με ένα κλάδο, πρέπει να λάβει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορούμε να συνομιλούμε με αυτούς που ε, φτιάχνουν το χρηματοδοτικό μέσο και λένε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, να μην μπορούν να λάβουν υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό το λένε όλοι. Και η συγχρηματοδότηση στο πρόγραμμα αυτό είναι αρκετά υψηλή γιατί είναι περίπου στο 40% κατά μέσο όρο. Θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη κατανομή. Ε, μπορεί να υπάρχει κατανομή σε κάποια μέτρα, αλλά μπορεί να είναι περισσότερη. Θα σταματήσω εδώ γιατί θα έχουμε και άλλε ευκαιρίες να τα συζητήσουμε. Κάτι ακόμα για τους δείκτες. Για τον προπολογισμό ε, τα ξέρουμε, αλλά ο κανονισμό λέει ότι πρέπει να έχουμε δείκτες. Αν δεν έχουμε δείκτε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θυμάστε ε, τη μάχη που δώσαμε μαζί Απ' τη μια έχουμε το παρατηρητήριο για τα οπτικοακουστικά μέσα που μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία ε, και δείκτες κλπ. Αλλά για την δημιουργική βιομηχανία δεν υπάρχουν δείκτες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ε, θέσουμε σοβαρά. Το Κοινό Κέντρο Έρευνας, το JRC, που εργάζεται, έχει τον προπολογισμό του κλπ. Δεν θα μπορούσε να έχει μια συγκεκριμένη δράση γι' αυτό να τους αναθέσουμε αυτό. Χωρίς να αρχίσουμε να λέμε και πάλι πρέπει να βρούμε επιπλέον πόρους κλπ. Δεν μπορούμε να αναθέσουμε μια αποστολή σε κάποιον ο οποίος ήδη υπάρχει. Έχουμε χιλιάδες ερευνητών που τώρα πια κάνουν και έρευνες και για τη δημιουργική βιομηχανία κλπ. Τέλο πάντων μπορεί να σας έχω και επιβαρύνει με όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ο κύριος Μόρκανο κάτι θέλει να πει. Μία ερώτηση μόνο. Από τη μία δείκτες, από την άλλη αξιολόγηση. Είναι δύο κεντρικά στοιχεία. Υπάρχουν και άλλα θέματα βέβαια. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Έχω αμφιβολίες, σέβομαι βέβαια τη δουλειά που κάνουν οι εκτιμητές εξ οι αξιολογητές εξ αλλά έχω και αμφιβολίες για το αν είναι σε θέση να εκφραστούν αντικειμενικά. Υπάρχει μεγάλη υποκειμενικότητα, υπάρχουν διαδικασίες που είναι λίγο μη διαφανείς. Σύντομα. Ο συνάδελφος ίσως από την ΑΣΕΑ θα μπορέσει να δώσει κάποιες απαντήσεις σχετικά με τις εγγύσεις. Το Σεπτέμβριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο θα μπορέσουμε να περιγράψουμε συστηματικά τις τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του οργάνου αυτού στην αγορά. Αλλά να πω γενικά ότι το θέμα αυτό καθορίζεται εν πολλής από τις αγορές. Ακριβώς επειδή δημοσιεύει και ασχολείται με τόσους πολλούς τομείς, Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο πολιτιστικό κομμάτι, στο οπτικοακουστικό κομμάτι, στην αρχιτεκτονική, τη μουσική, τα video games. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς τους ε, τραπεζίτες το τι θα κάνουν στον κάθε ένα από αυτόν τον τομέα. Δεν είναι σωστό. Η ιδέα είναι να τους βοηθήσουμε, να τους ενθαρρύνουμε αν θέλετε, να τους πούμε ότι θα μοιραστούμε κάποιους από τους κινδύνους μαζί σας, αλλά εσείς σαν επαγγελματίες έχετε σαν στόχο να ε, ορίσετε τα ε, δανειοδοτικά μέσα με όρους διαφορετικούς από την αγορά. Αυτό πρέπει να γίνεται σταδιακά, είναι η πρώτη φορά που το ξεκινάμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προκαταλάβουμε σήμερα. Η ευελιξία είναι η βασική λέξη εδώ. Διαφορετικά μέσα θα γίνονται διαθέσιμα από τις τράπεζες ανάλογα με το ε, πρόγραμμα το οποίο έχουν μπροστά τους. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Για το ΕΦΣΥ παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την αντίδραση των τραπεζών και των τελικών χρηστών, αυτών που ωφελούνται των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη γενικά του ΕΦΣΥ. Θα δούμε τι δυνατότητα θα υπάρχει μεταφοράς από το ΕΦΣΥ στο δικό μας μέσο αν πάει καλά το ΕΦΣΥ. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή, είναι δυνατόν δηλαδή να προβλεφθεί κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και από πλευράς του Και τέλος, σχετικά με τους δείκτες, θα πρέπει να κάνουμε την διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχουν από τη μία τα κριτήρια του κανονισμού, η νομική βάση που ορίζει τα τυπικά αν θέλετε κριτήρια αξιολόγησης και είναι χρήσιμα, θέλουμε να τα εμπλουτίσουμε όμως. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με τους ανεξάρτητους αξιολογιστές οι οποίοι κάνουν την ενδιάμεση λεγόμενη αξιολόγηση θα τους δώσουμε την δυνατότητα να προχωρήσουν στο έργο τους και μετά θα συζητήσουμε το θέμα με όλους τους εμπλεκομένους. Υπάρχει μια διαδικασία λοιπόν η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Για τα κριτήρια και τους εμπειρογνώμονες θα απαντήσει ίσως ο συνάδελφος από τη Νέα ΣΕΑ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, διαδικασία αυτή, την ότι καλά θα κάναμε να κοιτάξουμε και να συνεχίσουμε τη συνεργασία και με τα γραφεία που γνωρίζουν καλύτερα τους υποψηφίους και γνωρίζουν λοιπόν καλύτερα τι να γίνεται, αλλά και μαζί από τους, με τους εμπειρογνώμονες που είναι οι πελάτες, γιατί οι πελάτες είναι αυτοί που, οι εμπειρογνώμονες είναι αυτοί που διαβάζουν τις ε, ε αιτήσει και προσπαθούν να καταλάβουν σε τι βαθμό εξυπηρετούν του στόχου του προγράμματο. Και άρα, σε ό,τι αφορά ε, τι συζητήσει, θα μπορούσαμε να τι περιορίσουμε στο ελάχιστο σε ό,τι αφορά την εξελόγηση. Σε ό,τι αφορά του εμπειρογνώμονε, να θυμόμαστε ότι το βασικό καθήκον που επιτελούν οι εμπειρογνώμονε είναι μεμονωμένε αξιολογήσει, οι οποίε θα πρέπει να γίνονται βάσει όλων των πληροφοριών που ε, περιλαμβάνονται στην αίτηση. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και αυτό αποτελεί και ένα από τα βασικά παράπονα ε, των ε, υποβάλλοντων αίτηση των ετούντων. Ότι δεν κοιτάξαμε καλά δηλαδή την πρότασή του, το website του κτλ. Άρα θα πρέπει λοιπόν να γίνεται σωστή ανάλυση και εδώ μπορεί να βοηθούν οι εμπειρογνώμονε. Και αυτό μπορεί να γίνεται και εξ Δεν υπάρχει λόγο να είναι κανείς στο γραφείο. Γιατί όταν είναι οι εμπειρογνώμονες στο γραφείο, στην φάση αυτή τους λέμε να μην έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, να μην υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Το καλύτερο είναι όταν έχουν σχηματίσει ήδη μία άποψη, μετά να το συζητούν με τους ε, συναδέλφους τους για να μπορούν να συνενώσουν αυτές τις διαφορετικές τοποθετήσει και να συζητούν τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε την ε, Αναθεώρησε και την έρευνα αυτή και την ρωτάμε και την άποψη των εμπρευνομόνων. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι η πραγματική διαφάνεια είναι κοινή συζήτηση. Υπάρχει πρόβλημα και διαφάνεια κατά με. Σίγουρα θα ακούσουμε δηλώσει, περί μη σύγκρουση συμφερόντων κλπ. Αλλά νομίζω ότι σε αυτά τα πράγματα, αν όπω συνέβαινε νωρίτερα, που καθόμασταν όλοι γύρω από ένα τραπέζι και κινόταν μια συζήτηση, Πρέπει να υπάρχει λοιπόν κάτι πιο απτό και να υπάρχει και ένα κίνητρο. Να υπάρχουν και κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την κάθε χώρα, διότι υπάρχουν ε, κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Μπορεί να υπάρχει αμφιβολία ότι κανένας δεν κατάφερε να δει τίποτα. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην έχουμε αυτούς που πρέπει εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ένα πλαίσιο πίσω από την ζήτηση. Πρέπει λοιπόν να σας ευχαριστήσω που απαντήσατε και ειλικρινά όπως είπατε. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ο πρώτος σταθμός στην εκθεσή μας. Εγώ τουλάχιστον αυτό θεωρώ ότι είναι γιατί συγκεκριμένη ημέρα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή αλλά έτσι έχουν τα πράγματα στη ζωή. Θα κάνουμε το εξή λοιπόν. Πρώτον θα ξεκουραστούμε. Δεν ξέρετε εσείς, τι θα κάνετε. Εγώ πάντως ξέρω, κλείνουμε, να ευχηθούμε για καλό καλοκαίρι. Από τις 5 Σεπτεμβρίου όμως. Στη συνεδρία σε αυτή που θα είναι το απόγευμα και είστε όλοι προσκεκλημένοι, θα κάνουμε το δεύτερο επεισόδιο, θα γίνει και η παρουσίαση των εκθέσεων εγώ ποτέ δεν μου άρεσε να έχω και μαθήματα για το καλοκαίρι, αλλά αν θέλει κάποιο να ρίξει μια ματιά στα όσα σα διανύμαμε στα εγγραφά μα, να ευχαριστήσω και του συντάκτε των εγγράφων. Νομίζω ότι μπορεί να έχουν κάποια επιπλέον στοιχεία από αυτά που διαθέτουμε και να ξανασυζητήσουμε τότε. Και να έχουμε από εκεί και πέρα, εγώ τουλάχιστον θα ξεκινήσω, θα έχω πιο σαφείς ιδέες και θα έχω ακούσει και τους συναδέλφους που σήμερα δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες για να σας παρουσιάσω και το σχέδιο κειμένου μου. Φυσικά θα μπω στον κόπο να συναντηθώ με τους κοιόδης συζητητές πριν παρουσιάσω το σχέδιο κειμένου. Να ευχηθώ σε όλους. Ε, όποιος πρέπει ακόμα να μείνει στη δουλειά, ελπίζω να δουλέψετε για λίγο ακόμα. Όσοι πάτε διακοπές, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας από την Ευρωπαϊκή, όλους εσάς ε, και τους ευρωβουλευτές μας, τους παρόντες, τους απόντες, τη γραμματεία και φυσικά και τους διερμενείς που μας είναι απαραίτητοι. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Μιλήσαμε και για την πολυγλωσία σήμερα, οπότε ταυτιστήκατε κι εσείς με το θέμα που συζητήσαμε. Χίλια ευχαριστώ και ευχές σε όλους. Και κάτι ακόμα, συγγνώμη είχα λάβει τη δέσμευση με τον εαυτό μου να το πω. Ξέρω ότι είναι λυπηρό, αλλά δυστυχώ έτσι έχει ζωή. Προχθέ ε, χάθηκε ένα άνθρωπο που ήταν ε, αναπόσπαστο σημείο τη Δημιουργική Ευρώπη. Ένα νέο μουσικό, Ιταλός, ο Λορέντσο Αμούρι, που πριν από 20 χρόνια είχε ένα τύχημα στο σκι, ήταν πάρα πολύ καλός μουσικός και δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει πλέον τα πόδια και τα χέρια του, δεν μπόρεσε λοιπόν να κάνει μουσική και άρχισε να γράφει. Και πέρσι, φανταστείτε, κέρδισε το βραβείο Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας για την Ιταλία. Με ένα πολύ όμορφο βιβλίο που ανέφερε λίγο τη βιογραφία του. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω ότι με συγκίνησε γιατί πέρσι είχα την ευκαιρία να το απονείμω αυτό το βραβείο. Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί γιατί ήταν ήδη άρρωστος και ε, τον ε, άκουσε στο τηλέφωνο, ήταν ενθουσιασμένος και τον εξέπληξε που έλαβε ένα βραβείο που για πολλούς νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες έχει μια μεγάλη σημασία. Η Δημιουργική Ευρώπη λοιπόν είναι και αυτά τα πράγματα. Και στα πλαίσια τη Δημιουργική Ευρώπη υπάρχουν ε, και οι πολιτιστικέ πρωτεύουσε που συζητήσαμε, αλλά και τα βραβεία, όπω για παράδειγμα το λογοτεχνικό βραβείο. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λοιπόν με μια ε, ανάμνηση αυτού του ανθρώπου που εκπροσωπούν του καλλιτέχνε, αυτού του δημιουργού που και χωρί δείκτε αξίζει τον κόπο να γνωρίσουμε στη ζωή. Ευχαριστώ πολύ.